Είναι η ώρα 3. Και είμαστε και τρεις μόνο μες στην αίθουσα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε ελεκτικό συνέδριο. Καλώς ήρθατε κυρία Επίτροπε και λοιπή Επιτροπή. Θα προσπαθήσω να διαβάσω το όνομά σας. Κιόκαν Κουίν, καλά τα λέω. Θα το έχω μάλλον κατακριουργήσει, αλλά ξέρετε ότι έχουμε και ένα κοινό σημείο ότι και εσείς και εγώ είμαστε υπήκοοι χώρας άνευ κυβερνήσεως. Δεν ξέρω αν αυτό είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα. Πάντως στη χώρα μου το ότι δεν υπήρχε ε, κυβέρνηση απέβησε καλό για την Ευρώπη. Είναι το σύστημα των των δοχείων. Βρισκόμαστε εδώ λοιπόν με μια διαδικασία απαλλαγής, πολύ σημαντική. θέματα και δική σας αρμοδιότητας. Και πάντα προσπαθούμε βέβαια να σας βλέπουμε εδώ, να συζητούμε με βάση την κοινή λογική, με γνώμονα την κοινή λογική να καταλήγουμε σε συμπεράσματα. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Νόακ να μας πει τι γνώμη έχει για όλα αυτά. Ο ίδιος και η συνεργάτες του, μετά στην ε, κυρία Επίτροπη και βέβαια και στον κύριο Συγητή. Με την ελπίδα ότι θα έρθουν ε, οι συνάδελφοι συν και εγκαίρως. Ο κύριος Νόακ έχει το λόγο από το ελεγκτικό συνέδριο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, κυρία Επίτροπε, κύριε Μόιλε, θέλω να πω, είναι η δεύτερη και μάλλον τελευταία φορά είναι η τρίτη και μάλλον τελευταία φορά που παρουσιάζω στην Επιτροπή σας τα συμπεράσματα του ελεγκτικού συνεδρίου στους τομείς πολιτικής της Ερευνά τη ε, Κοινωνία τη Πληροφορία των μεταφορών της ενέργειας, στο πλαίσιο της ε, δηλώσεω συμμορφώσεως. Και αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι πλέον αναλαμβάνω καθήκοντα για τα ε, ταμεία συνοχής, για τα οποία θα σα παρουσιάσω του χρόνου τα σχετικά συμπεράσματα. Έτσι λοιπόν, η δαπάνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση του ε, πολιτικής πολιτική ανέρχεται σε 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009, δηλαδή 7,5% των συνολικών δαπανών τη Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009. Στο κεφάλαιο 5 των αιτήσεων τη ετησία εκθέσή μα, επικεντρωνόμαστε κυρίω σε δαπάνε έρευνα και πρέπει να σημειώσουμε ότι στο είναι ομάδα πολιτικής, στο σύνολό τη ε, βλέπουμε ότι 70% των κονδυλίων ε, αφιερώνονται από τις δαπάνες σε ερευνητικά προγράμματα υπό το πολιετέ ε, πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Τα πολιετή μάλλον προγράμματα. Και έχουμε πάνω από 12.000 δικαιούχου, εκ των οποίων 250 μεγαλύτεροι έχουν εισπράξει το 5% περίπου της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την έρευνα. Η προσεχής κατηγορία δαπανών είναι αυτή της ενέργειας και των μεταφορών, των σχετικών σχεδίων δηλαδή, που αναπτύσσονται υπό το πρόγραμμα των διευρωπαϊκών δικτύων. Το μεγαλύτερο τμήμα των δαπανών αυτής της ομάδας ε, πολιτικής ε, τίθεται υπό τη διαχείριση απευθείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τι όλο και περισσότερο παρεμβαίνουν εκτελεστικές ε, υπηρεσίες και κοινέ δράσεις. Ω εκ τούτου, η πλειονότηση των πληρωμών που δειγματοληπτικά ελέγχθησαν από το ελεγκτικό συνέδριο έχουν να κάνουν με τα προγράμματα πλαίσιο, ιδιαίτερα στα ενδιάμεσα και τελικά, τα ενδιάμεσα και τελικά ποσά πληρωμή ε, για το πρόγραμμα πλαίσιο υπαριθμών 6 και τις προκαταβολές για το υπαριθμών 7. Ο κύριος κίνδυνος ως πω, στην νομιμότητα και την ε, ε, κανονικότητα των δαπανών στον τομέα της έρευνας είναι να ε, υπερβάλλει ο δικαιούχος το κόστος που υποβάλλει προς έγκριση στις δηλώσεις του ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στις δηλώσεις ιδιαίτερως για αποζημίωση δαπανών. Εάν αυτό δηλαδή δεν προληφθεί, δεν διαγνωστεί, δεν διορθωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει πρόβλημα. Το 2009 λοιπόν έλεγξε το συνέδριο ένα δείγμα 150 πληρωμών και αξιολόγησε τους, ε, τα συστήματα ελέγχου, ιδιαίτερα ως προς τις πληρωμές στην έρευνα, συμπεριλαμβανομένης και της πρόοδου στην εφαρμογή της ε, εκ των εξτέρων ε, λειτουργίας ε, δημοσιονομικού ελέγχου και στρατηγικής δημοσιονομικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι δείχνουν λοιπόν αυτά τα, αυτή η έλεγχη. Τα αποτελέσματα του 2009 στους δημοσιονομικούς ελέγχους επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τα πορίσματα των προηγούμενων δύο ετών, δηλαδή είχαμε εκτιμήσει πιθανό ε, ποσοστό σφάλματος μεταξύ 2 και 5% και μάλιστα μάλλον χαμηλό, δηλαδή πιο κοντά στο 2 παρά στο 5%. Ε, λοιπόν το συνέδριο ότι 36 από 36 ή 24% από τις συναλλαγές που έχουν ελεγχθεί ε, είχαν ε, κάποιο πρόβλημα, σφάλμα δηλαδή. Στις 23 περιπτώσεις πρόκειται για ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές, ελεγκτικά προγράμματα, σχέδια του ε, προγράμματος πλαισίου 6 και του 7. Οι δε δραστηριότητες επιπτίας και ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν εν μέρη αποτελεσματικές ως προς την εξασφάλιση της του εύρυθμου των πληρωμών. Αναγνωρίζει το Ελεκτικό Συνέδριο, δε, όπως και πέρσι, ότι οι προσπάθειες που κατέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση των ελεκτικών συστημάτων και για την απλούστευση ε, του τρόπου χορήγηση των κονδυλίων είναι ουσιαστικές και αυτό ταυτόχρονα εξηγεί τη μειωτική τάση στο ποσοστό σφάλματος, ωστόσο δεν εξασφαλίζει ότι θα συνεχιστεί και στο πρόγραμμα πλαίσιο παριθμών 7 και στα λοιπά προγράμματα πλαίσια η ίδια αυτή τάση και υπάρχουν ακόμη κίνδυνοι να, ε, να επαναληφθούν προβλήματα που είχαμε δει ήδη στο 2009. Επιτρέψτε μου λοιπόν να εξηγήσω τα κύρια συμπεράσματά μας. Η κύρια πηγή σφάλματος έχει να κάνει με την επιστροφή υπερβολικών δαπανών είτε προσωπικών είτε έμεσων. Ε, για το 2008 τα περισσότερα από αυτά τα σφάλματα είχαν να κάνουν με τις ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές σε δικαιούχους προγραμμάτων συμβάσεων καλύτερα ε, ερευνητικών που είχαν ε, υποβάλει δηλώσεις δαπανών συχνά συνοδευόμενες και από πιστοποιητικό δημοσιονομικού ελέγχου και είδαμε σφάλματα και για το πρόγραμμα πλαίσιο 7 όπως και για το 6. Εντοπίζουμε λοιπόν τα εξής, ότι πώς προβλέπονταν έφεραν καρπούς ή εκ των προτέρων ε, εξ αποστάσεως έλεγχοι με λίγες εξαιρέσεις που μπορούν να περιοριστούν ε, εάν διαγνωστεί εγκαίρος το σφάλμα και αντισταθμιστεί από άλλους τύπους ελέγχου. Δεύτερον, τα πιστοποιητικά δημοσιονομικής συμμόρφωσης δεν προσφέρουν επαρκή ασφάλεια ακόμη και το σχετικό επίπεδο σφάλματος με πιστοποίηση, δηλαδή δημοσιονομική πιστοποίηση στο κόστος, στις δηλώσεις κόστους ήταν ίδιο, ίδιο με το περσινό, δηλαδή 43%. Και ενώ τρίτον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσπαθήσει να εξαπλουστεύσει την ε, διαδικασία ε, πιστοποίησης δημοσιονομικού ελέγχου υπό το πρόγραμμα πλαίσιο υπαριθμών 7 με την ε, εκ των προτέρων πιστοποίηση του τρόπου κοστολόγησης του δικαιούχου. Το συνέδριο διαπιστώνει ότι το σύστημα δεν μπόρεσε να φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα τουλάχιστον ακόμη και στα τέλη του Μαΐου του 2010 μόνο 25 από τους δυνάμει 650 ε, δικαιούχους είχαν λάβει την εκ των προτέρων πιστοποίηση των μεθοδολογιών κοστολόγησης που ακολουθούν. Έτσι, μεγάλοι δικαιούχοι ε, φαίνεται να προτιμούν την εφαρμογή Φαίνεται μάλλον να μην ε, προτιμούν την εφαρμογή αυτής της μεθόδου ισχυριζόμενοι ότι δεν ε, ευθυγραμμίζεται με τις κοινέ λογιστικές πρακτικές που εφαρμόζουν στο εσωτερικό της, ε, ε, χώρο τους και γενικά στις ερευνητικές δραστηριότητες. Αυτό έχει μια κάποια ευστοχή ως επιχείρημα και ίσως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ταυτόχρονα Υπαριθμών 4 εντοπίζουμε ορισμένες θετικές εξελίξεις ως προς την στρατηγική εκ των υστέρων δημοσιονομικών ελέγχων στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου υπαριθμών 6. Δηλαδή, η επιτροπή δηλαδή, επιτροπή δηλαδή εξασφαλίζει τους στόχους της ως προς τους ελέγχους για την ε, χρονιά ολόκληρη και συνεχίζει τις προσπάθειές Πιστεύουμε ότι αντίστοιχα έχουν ξεκινήσει οι δημοσιονομικοί έλεγχοι και υπό την ε, στρατηγική δημοσιονομικού ελέγχου στο πρόγραμμα πλαίσιο υπαριθμών 7 η ανάκτηση και η δημοσιονομική διόρθωση ε, στη συνέχεια βλέπουμε ότι ενισχύονται αλλά παραμένουν ακόμη και μάλιστα ενισχύονται ταυτόχρονα και τα μη ανακτηθέντα ποσά. Επίσης σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι το 2009 η Επιτροπή ξεκινάει την εφαρμογή ενός μηχανισμού κυρώσεων που ήδη προβλέπεται το πρόγραμμα πλαίσιο 6. Εν τέλει το ελεγκτικό συνέδριο διαπιστώνει ότι η δηλώσεις, αιτήσεις δηλώσεις δραστηριοτήτων και οι δηλώσεις ε, των γενικών διευθυντών, ε, των γενικών διευθύνσεων για την έρευνα, τα δημοσιονομικά, τα διευρωπαϊκά δίκτυα και την κοινωνία της πληροφορίας δίνουν μια ικανοποιητική αξιολόγηση της δημοσιονομικής διαχείρισης σε σχέση με την κανονικότητα των λογαριασμών και φτάνω τώρα στα συμπεράσματα για να ε, πω ότι δεν μπορούμε παρά να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει προσπάθειές της ως προς την εξασφάλιση ενός αυστηρού, μιας αυστηρής ε, ε, εφαρμογής των αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου, ιδιαίτερως εξασφαλίζοντας ότι οι δημοσιονομικές αρχές αρμόδιες για την πιστοποίηση θα είναι εν γνώση των κριτηρίων επιλεξιμότητας μέσω της αναθεώρησης της λειτουργίας του συστήματος για την πιστοποίηση και των ε, μεθόδων κοστολόγησης των δικαιούχων προκειμένου να περιοριστεί η καθυστέρηση η βραδιπορία δηλαδή στις ανακτήσεις και προκειμένου να επιβληθούν εφόσον χρειάζεται κάτι τέτοιο και κυρώσεις. Επιπλέον ε, σημειώνουμε ότι υπάρχει περιθώριο για βελτίωση και απλούστευση των όρων χρηματοδότηση τη έρευνα ε, και ιδιαίτερα τα, θεωρούμε τα μέτρα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στο θέμα αυτό. Η απλούστευση και η διευκρίνηση των κανόνων είναι πολύ σημαντική και για την κανονικότητα των δαπανών. Αποτελούν δε βασικό μέσο για την επίτευξη των ευρωπαϊκών πολιτικών στοχεύσεων. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη σύνοψη. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Επίτροπο. Τι έχετε να απαντήσετε στα όσα μας είπανε. Κύριε Στάες, κύριε Αντιπρόεδρε, αξιόπτημα μέλη, δόκτωρα Νόακ, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι εδώ ως Ευρωπαία Επίτροπος για την έρευνα και την επιστήμη και θα ήθελα να ε, σας πω ότι η καλή χρηματοδότηση για την έρευνα είναι μία από τις βασικές μου προτεραιότητες. Σήμερα είμαι εδώ για να απαντήσω στις παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2009 και να απαντήσω στις ερωτήσεις των μελών για την έκθεση αυτή. Καταρχάς ε, θα ήθελα να σας πω ότι δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έχουμε κάνει και εμείς μια αντίστοιχη ανάλυση και η ειδική ως μας ο έλεγχος καταδεικνύει αντίστοιχα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα που επιτύχαμε μέχρι τούδε και που ε, αναγνωρίστηκαν συγκεκριμένα από το ελεγκτικό συνέδριο στην έκθεσή τους και από τον κύριο Νόακ ε, σήμερα είναι πολύ καλά. Έχουν μειωθεί τα αρνητικά μας στοιχεία τα τελευταία χρόνια και παρά το γεγονός ότι το συνέδριο αναγνωρίζει ότι έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις υπάρχουν κάποιες ελλείψεις τις οποίες θα πρέπει ακόμα να αντιμετωπίσουμε. Οι ανησυχίες ε, μας είναι για την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των πιστοποιητικών ελέγχου, ε, έλεγχη για τους δικαιούχους, ε, μέσο κόστος για το προσωπικό και μείωση των καθυστερήσεων για την ανάκτηση ποσών τα οποία καταβλήθηκαν όταν επιβλήθηκαν κυρώσεις. Όσον αφορά στα πιστοποιητικά, θα πρέπει καταρχάς να υπενθυμίσουμε ότι το θέμα αυτό αφορά κυρίως το πρόγραμμα πλαίσιο 6 η ανάγκη να υπάρχουν επιστοποιητικά ελέγχου έχει μειωθεί σημαντικά στο πρόγραμμα πλαίσιο 7 για να μειωθεί το γραφειοκρατικό έκθος για τους δικαιούχους όταν υπάρχουν ακόμα πιστοποιητικά ελέγχου έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των πιστοποιητικών που εκδίδονται από εξωτερικούς ελεγκτές. Επίσης αναγνωρίζεται ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η διαδικασία του ε, προγράμματος πλαίσιο 7 για να χρησιμοποιήσουμε και τις μεθοδολογίες για τους δικαιούχους για να δούμε τι γίνεται με τα κονδύλια. Επίσης αυτό λαμβάνει υπόψη και τη δική σας τη σύσταση για να μειώσουμε το κόστος για το προσωπικό και να έχουμε μεθοδολογίες οι οποίες συνάδουν με τις τρέχουσες επιχειρηματικές πρακτικές. Εχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υιοθέτησε μία ανακοίνωση για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα πλούστευσης, τα οποία αναγνωρίζει ότι ε, δεχόμαστε εν γέννη τις μεθοδολογίες μέσου υπολογισμού προσωπικού για τις τρέχουσες πρακτικές και μπορούμε να δούμε το τρέχον κόστος για το προσωπικό όπως καταγράφεται στις επιχειρήσεις. Το συνέδριο αναγνωρίζει ότι ο αριθμός των μη επιλέξιμων δαπανών τα οποία, ο, οι οποίες ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2009 αυξήθηκε και έχουν επιβληθεί και ανάλογες κυρώσεις. Αλλά τα ποσά τα οποία ανακτήθηκαν και κυρίως ε, κάποιες ε, περιπτώσεις προβολών είναι ακόμα λόγος ανησυχίας και τα μέτρα τα οποία εισαγάγαμε το Δεκέμβριο του 2009 θεωρούμε ότι θα απλουστεύσουν και θα επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία. Αυτές είναι λοιπόν οι δράσει οι οποίε αναλάβαμε για να ανταποκριθούμε στι συγκεκριμένε συστάσεις που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Επιτρέψτε μου τώρα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις όσον αφορά την ε, καλή οικονομική διαχείριση και τη χρηματοδότηση και την ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης, ελέγχου και τα ωφέλεια ε, για το κόστος ε, από τους ελέγχους εφαρμόστηκε μία αυστηρή πολιτική ελέγχων που στόχο είχε να μειώσει το ποσοστό σφαλμάτων στο 2% που εφαρμόζεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αλλά φυσικά υπάρχει και ένα ατίμημα. Συγκεκριμένα ε, η ανθρώπινη και οικονομική πόρη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τους δικαιούχους ε, ήταν ε, απαραίτητη και υπήρχαν πολλές διαμαρτυρίες από την επιχειρηματική κοινότητα αλλά και την επιστημονική κοινότητα για το υπερβολικό άχθος. Ο βασικό μα στόχο θα πρέπει λοιπόν να είναι να απλουστεύσουμε ακόμα περισσότερο τη χρηματοδότηση για την έρευνα. Όπως ε, ε, μα υποδείχθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο και επαναλήφθηκε και σήμερα από τον καθηγητό ε, την ΟΑΚ, οι απλουστευμένε διαδικασίε είναι η καλύτερη διασφάλιση τη μείωση των ποσοστών σφαλμάτων και συμφωνούμε όλοι από αυτού. Δεν θα πρέπει λοιπόν να έχετε καμία αμφιβολία για το γεγονό ότι εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι πρέπει να προχωρήσουμε με την απλούστευση. Μόλις ανέλαβα καθήκοντα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια διαδικασία για απλούστευση των προγραμμάτων έρευνας και μας επιτρέπει να έχουμε πολύ σημαντική απλούστευση βάσει του τρέχοντος προγράμματος πλαίσιο, η οποία θα εφαρμοστεί ε, βάσει μιας απόφασης που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εχθές. Θα έχουμε ε, υπολογισμό του μέσου κόστους και το προσωπικό και θα γίνεται, υπάρχει δυνατότητα να αποζημιώνονται όλα τα μέλη ε, των επιχειρήσεων από τις flash rate πληρωμές. Επίσης όλα αυτά περιλαμβάνονται στην ε, τριετή αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού τα μέτρα αυτά ε, συνάδουν με τα όσα πρότεινε η έκθεση Καρβάγιο για την ε, απλούστευση που ενέκρινε ε, το Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο. Θα μπορέσουμε να προτείνουμε πιο ριζοσπαστικέ απλουστευμένες διαδικασίες στο επόμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης επί τη βάση και της προτινόμενης αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση Καρβάλιο. Χρειαζόμαστε λοιπόν την υποστήριξη των θεσμικών οργάνων και του Κοινοβουλίου φυσικά για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Παρά το γεγονό ότι η απλούστευση των μελλοντικών προγραμμάτων που θα βασίζεται σε απλούστερου δημοσιονομικού κανόνε είναι ο βασικό μα στόχο, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι επιπτώσει του τρέχοντο πιο περίπλοκο συστήματο κανόνων, δυστυχώ θα πρέπει να μα ακολουθήσουν για χρόνια. Οι τρέχοντε κανόνε για το πρόγραμμα πλαίσιο 7 θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι το 2017 και ίσω και αργότερα. Τα μέτρα τα οποία εγκρίναμε χθε μπορεί να μειώσουν τα σφάλματα, αλλά κάποια άλλα μέτρα για του εκ των προτέρων ελέγχου ε, στο πρόγραμμα πλαίσιο 7 μπορεί να αυξήσουν τα ε, προβλήματα σε σχέση με το πρόγραμμα πλαίσιο 6. Έτσι, μπορεί τα αρχικά σφάλματα στο πρόγραμμα πλαίσιο 7 να μην αποκλίνουν ουσιαστικά από το πρόγραμμα πλαίσιο 6. Αυτό σημαίνει ότι ε, δεν, θα πρέπει να, δεν σημαίνει συγγνώμη, ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε την ίδια στρατηγική ελέγχου με το πρόγραμμα πλαίσιο 6. Και τι είναι το, ποιο είναι το όφελο για το πρόγραμμά μα. Θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε του καλύτερου ερευνητέ παγκοσμίω και να μπορέσουμε να ε, πείσουμε του επιχειρηματίε, τα πανεπιστήμια και άλλε ερευνητικέ ε, μονάδε ε, για την Ευρώπη ώστε να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε και ελπίζω η το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απλούστευση των ερευνητικών προγραμμάτων ε, να υποστηρίζει πλέον την αποδοχή ενός ε, ανεκτού επίπεδου ε, σφαλμάτων για τα ερευνητικά προγράμματα. Ανεκτό σημαίνει μεταξύ του 2 και του 5% που σημαίνει ότι θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει τη στρατηγική ελέγχου της και να εστιάσει περισσότερο σε στοχευσμένους ελέγχους που θα βασίζονται στον κίνδυνο και να κάνει συγκεκριμένου αυξημένους παρά να δαπανεί τεράστια ε, κονδύλια ε, για τους ελέγχους για την έρευνα. Ο κίνδυνος σφάλματος δεν σημαίνει ότι θα έχουμε αυτόματα κυρώσεις μόλις διαπιστώνονται σφάλματα. Η αρχή θα είναι ότι θα ανακτώνται όλα τα υπερβολικά κονδύλια και όπως σας εξήγησα πριν, αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε τις προσπάθειες να μειώσουμε τα σφάλματα ακόμα περαιτέρω στα μελλοντικά προγράμματα και να έχουμε και πιο απλουστευμένους κανονισμούς και κανόνες και διαδικασίες και να καταλήξουμε σε ένα ε, κατόφλι του 2% ή ακόμα λιγότερο ή δυνατόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον εισηγητή. Ο κύριος Χατζημαρκάκης είναι ο βασικός εισηγητής και στη συνέχεια θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε μια αρχή ping-pong, ε, απάντηση και ερώτηση απευθείας. Δεν ξέρω ποιος θέλει να παρέμβει από τις συναδέλφους. Ε, σας παρακαλώ, πέστε μου για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με ένα κατάλογο αγορητών. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη γραπτή απάντηση στα γραπτώς υποβληθέντα ερωτήματα. Προκύπτει βέβαια μια σειρά από που έχουν να κάνουν με τη ε, δυνατότητα βελτίωση των μελλοντικών μας εργασιών. Θα ήθελα να συνεχίσω στα όσα είπε ο Δ. Νόακ ως προς τα κύρια σημεία επικρίσεως και να αναφερθώ στην... Ε, σε ορισμένα σημεία ως προς την, ε, τους δημοσιονομικές διορθώσεις καταρχάς, δηλαδή γιατί το κενό μεταξύ των όσων ε, κακώς κατεβλήθησαν και των ανακτηθέντων ποσό, ποσών όλο και μεγαλώνει. Επίσης θα θέλω να φερθώ και στο ανεκτό ή αποδεκτό ε, τον αποδεκτό κίνδυνο σφάλματος και να δούμε λίγο και τα συγκεκριμένα αριθμητικά. Τώρα, σαν αφορά τη δημοσιονομική διόρθωση. Διαπιστώνει το ελεκτικό συνέδριο ότι εκ των προτέρων έλεγχη σε εσά είναι άμεμπτοι, είναι ελάχιστα τα προβλήματα, μπορούμε και μόνο να σας ε, ε, συγχαρούμε γι' αυτό. Είναι καταπληκτικό δηλαδή αυτό το κομμάτι που αφορά τον έλεγχο των δραστηριοτήτων σας και ελπίζω να έχουμε το ίδιο, όπως άλλωστε βλέπουμε και γενικά στις λοιπές ε, γενικές διευθύνσεις. Έχει να κάνει με τις προκαταβολές λίγο πολύ αυτό. Όσον όμως αφορά τους εκ των υστέρων ελέγχους διαπιστώνονται κάποιες δυσκολίες οι οποίες συν το χρόνο ενισχύονται, αυξάνονται. Φυσικά αυτό σχετίζεται και με το γεγονός ότι έρχονται στην ε, τελική τους φάση όλο και περισσότερα προγράμματα του προγράμματος πλαισίου παριθμών 6 και άρα έρχεται η ώρα του ελέγχου καμπύλη που παρουσιάζει το ηλεκτρικό συνέδριο, αυτό το κενό δηλαδή, το, η ψαλίδα, έχει να κάνει και ιδιαίτερο με το γεγονός ότι έρχονται με καθυστέρηση οι πληρωμές. Όσο πιο καθυστερημένες λοιπόν είναι οι πληρωμές, τόσο πιο αργά έρχεται και η ολοκλήρωση το κλείσιμο των προγραμμάτων και τόσο πιο δύσκολο να επαληθευθεί και να ανακτηθεί καλύτερα το ποσό που ενδεχομένως έχει χρησιμοποιηθεί. καταβληθεί. Ερωτώ λοιπόν αυτή η ψαλίδα πώς την ε, ε, εξηγείτε και τι μπορείτε να κάνετε ώστε να περιοριστούν τα χρονικά περιθώρια. Να γίνεται αμέσως δηλαδή ο έλεγχος, χωρίς άλλη βραδιπορία. Αν μου επιτρέψετε θα δώσω όλες τις ερωτήσεις ε, ομού. Έχουμε λοιπόν επίσης το θέμα της απλούστευσης. Και εδώ εκφράζω την ικανοποίησή μου για το ότι και εσείς κύριε Επίτροπε Έχετε αποδειχθεί σε έναν πολύ εντατικό ε, διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά φερθήκατε και εσείς ρητά στην έκθεση Καβάλιο, όπου είχαμε και το θέμα της απλούστευσης ε, ε, ω κύριο ζήτημα και πρέπει να πω και στις ακροάσεις μας με τους επιτρόπους, με όλους τους επιτρόπους, ωραία λόγια, μεγάλα λόγια, όλοι ζητούν την απλούστευση. Όταν όμως έρχεται η ώρα της εφαρμογής αυτής, της υλοποίησης, εμείς ως βουλευτές Ίσως να ζητούμε κάπως περίπλοκους κανόνες, το παραδέχομαι, αλλά ίσως και να είναι και τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία πολύ συχνά ε, κρύβονται, φυλάγονται πίσω από πολύ περίπλοκους κανόνες με τις εθνικές φερρυπίν ε, υπηρεσίες υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων έρευνας που με χαρά βλέπουν ότι λίγοι καταλαβαίνουν τι συμβαίνει ε, με τους κανόνες αυτούς. Είναι κάτι σαν την Καθολική Εκκλησία στον ε, Μεσαίωνα που ε, έλεγε τη λειτουργία στα λατινικά για να μην καταλαβαίνει κανείς περί τίνος πρόκειται. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να αναπτυχθεί περισσότερο αυτό το πρόγραμμα δράσης. Η έκθεση Καρβάλιο ασφαλώς υποδεικνύει μια σωστή κατεύθυνση. Ερωτώ όμως κυρία Επίτροπε και εσείς συγκεκριμένα τι μπορείτε να μας πείτε ότι θα κάνετε προκειμένου τα αρνητικά παραδείγματα, τα κακά παραδείγματα που έχουν εντοπιστεί ε, να αντιμετωπιστούν και βέβαια στον δρόμο αυτό σας ακολουθήσουν και τα κράτη-μέλη. Χαίρομαι για τη διάθεση για καινοτομία, για ε, αλλαγή. Δεν πρόκειται για ένα καινούριο εργαλείο βεβαίω, αλλά για μια νέα τεχνική περισσότερο, ώστε ε, να γίνει το streamlining, όπως λέμε ωραία στα γερμανικά, των νέων προγραμμάτων ή των πολλαπλών προγραμμάτων. Υπάρχουν βέβαια διαφορετικά μέσα προωθησής ενίσχυσης ε, αλλά ίσως είναι και θέματα που ανήκουν περισσότερο στις αρμοδιότητε τη ΣΥΤΡΕ, τη επιτροπή δηλαδή Έρευνας. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία ίσως η τροποποίηση κάποιων ε, διατυπώσεων για την καταβολή των ποσών ε, να πρέπει να μας απασχολήσει ειδικότερα. Τα λάμψαμς, δηλαδή τα κατά αποκοπήν ποσά ιδιαιτέρως, ε, είναι πιο δύσκολο να υπολογιστούν. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι μπορεί κανείς να διευκολύνεται με την ε, καταβολή ενός καταποκοπήν ποσού εάν υπάρχει πολύ μεγάλος κατακαιρματισμός, αν πρέπει παραδείγματι να δίνουμε με λεπτομέρεια την κάθε ώρα ή ανθρωπόρα ως τρόπο υπολογισμού των δαπανών. Αλλά πρέπει να υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος και πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα της απλούστευσης αλλά και της συμπίεση ταυτόχρονα του κινδύνου σφάλματος. Καταλαβαίνω βέβαια το επιχείρημα που θα μου πείτε ότι το 2% σημαίνει υπερβολικά πολλές ε, διατάξεις, διατυπώσεις ασφαλείας προκειμένου να συμπιέζουμε τον κίνδυνο του σφάλματος το 2%. Και έχω κάνει και εγώ βέβαια τις ε, επισκέψεις μου, έχω δει επιτόπου πως ε, γίνεται η δουλειά σας και βλέπω ότι και στατιστικά ακόμα ε, όχι μόνο κοστίζει πολύ όλος αυτός ο έλεγχος, όλες αυτές οι διαδικασίες ε, που γίνονται οι πολλαπλές, αλλά ταυτόχρονα και οι ελέγχοντες, οι ελεγκτές καλύτερα, αισθάνονται μια κάποια ε, δυσαρέσκεια ψυχολογικά, αισθάνονται πίεση δηλαδή, γιατί διαρκώς έρχονται να επαναλάβουν τον ίδιο έλεγχο, τον ίδιο έλεγχο διαρκώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως θα πρέπει να δούμε διαφορετικά, αν όχι για το πρόγραμμα πλαίσιο 7, για το 8 πλέον. Αλλά θα ήθελα στην απάντησή σας να σας ρωτήσω το εξής. Όταν, ε, και αναφέρομαι ειδικά σε τομείς που έχουν πολλές, ε, έχουν αυξημένο κίνδυνο ή παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο. Γιατί δεν επικεντρώνεστε σε αυτούς ακριβώς τους τομείς. Πρώτα-πρώτα. Έτσι ώστε να αποκλείσετε τις χειρότερες περιπτώσεις από τη χρηματοδότηση. Και εδώ, το έχουμε ξανασυστήσει άλλωστε νομίζω, σας επιβεβαιώνω ότι η Επιτροπή μας έχει πολλούς δισταγμούς ως προς την αύξηση του επίπεδου αποδεκτού σφάλματος. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει περίπτωση στην έρευνα ο κίνδυνος να αυξάνεται, γιατί είναι πολύ πιο αφηρημένο το αντικείμενο. Έρευνα δεν σημαίνει, δε, η έρευνα είναι κάτι το πολύ πιο αφηρημένο και το πολύ πιο γενικό. Δεν είναι τόσο απτό όσο το να πούμε κατασκευάζω μια γέφυρα και κοστίζει τόσο, θα κοστίσει τόσο, έχει κοστίσει τόσο. Στην έρευνα ίσω είναι κάπω πιο, πιο σαφή τα πράγματα. Αλλά πάλι χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν πιο πολλέ αποδείξει και πιο μικρό ποσοστό σφάλματο. Και μια μικρή ερώτηση για τι ε, διατυπώσει ε, πληρωμή. Αυτή τη στιγμή προβλέπεται ότι ακόμη και ο ετών ο οποίος έχει δικαίωμα και έχει πάρει τη σχετική έγκριση θα εισπράξει τα χρήματα με ένα χρόνο καθυστέρηση, ένα χρόνο αργότερα. Αυτό είναι πάρα πολύ. Εάν ε, βάλουμε δε στο παράδειγμα μια μικρομεσαία επιχείρηση, μια μικρομεσαία, ένα μικρομεσαίο ερευνητικό κέντρο, προφανώς αυτή η καθυστέρηση προξενεί πολλές δυσκολίες. Και εδώ βέβαια θα το συνδυάσω και με το νέλεχο Επομένως και η προκαταβολή και οι έμεσες πληρωμές βλέπουμε ότι δεν έχουν τόσα προβλήματα όπως ε, ε, επισημαίνει και το ελεγκτικό συνέδριο. Στην τελική πληρωμή και το κλείσιμο και μεγάλη καθυστέρηση παρουσιάζεται και αντίστοιχα δυσκολία και καθυστέρηση στην ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων. Και επανέρχομαι με μια τελευταία παρατήρηση. Το πρόγραμμα πλαίσιο 7 έχει 55 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά ως πρικοδότηση. Νομίζω είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πρόγραμμα. Και σας λέω τίμια, έντιμα, ότι δυσκολεύομαι να εξηγήσω στον πολίτη και ψηφοφόρο μου τι προσφέρει αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο, αυτό το more value for money, πιο πολλά με τα λεφτά αυτά ή με τα λιγότερα λεφτά, τι σημαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι πολλοί οι δικαιούχοι οι οποίοι έχουν μπει στο σύστημα και υποφελούμενοι από δωρεές, δηλαδή ε, χορηγία η οποία δεν επιστρέφεται, ε, κάνουν τη δουλειά του, ενώ θα μπορούσαν ωραιότατα να δουλεύουν με, το σύστημα του δανείου, loan, με στροφή δηλαδή τελικά του κεφαλαίου. Και πιστεύω ότι εν προκειμένου είναι πάρα πολύ καλή ιδέα το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Ίδρυμα, όπου ασφαλώ χρειάζονται οι δωρεέ, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί κανεί να, να κάνει τη δουλειά την ερευνητική αν δεν υπάρχει δωρεά σε επίπεδο ε, Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Ιδρύματο. Αλλά πέραν αυτού, δεν μπορούμε να το βελτιώσουμε, δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των σχεδίων και την ορετότητά του για τον πολίτη. Μια και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο που να σκοπεύει να φέρει φερειπίν τον άνθρωπο στη σελήνη, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πιο ουσιαστικό και πιο πρακτικό. Ευχαριστώ. Ε, λοιπόν, τρεις έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Βανόβα, ο κ. Φιέλνερ ο κ. Σοντή και η κυρία Γιάλα Σέντερ. Δεν υπάρχει άλλος. Θα σας δώσω το λόγο για μία ακόμη φορά για να απαντήσετε στις ερωτήσεις του εισηγητού. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσω τις ερωτήσεις όσο πιο πλήρω γίνεται, χωρίς να μακρηγορώ, διότι έχετε περιορισμένο χρόνο. Όσον αφορά την ανάκτηση, ότι τα εκκρεμία ανακτήσιμα από τριπλασιάστηκαν σχεδόν το 2009. Αυτό δεν οφείλεται σε μία μείωση ρυθμού ανακτήσεων, αλλά λόγω της νέας ενισχυμένης στρατηγικής ελέγχου που εφαρμόστηκε 2007-2008. Λοιπόν, στρατηγική για το πρόγραμμα πλαίσιο μας επέτρεψε να εντοπίσουμε μη επιλέξιμο κόστος και να το ερευνήσουμε κατά συμμετέχοντα σε πρόγραμμα σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι κατά παρελθόντα έτη. Για το πρόγραμμα πλαίσιο 6, το ανακτήσιμο ποσό έπαψε να αυξάνεται το, 2000, το τέλος του 2010 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, μάλλον η προσπάθεια ανάκτησης έχει πάρει μια ορμή και το σημαντικότερο ποσό της ανακτήσεως του προγράμματος πλαισίου 6 θα ολοκληρωθεί μάλλον τον επόμενο χρόνο και το μεγαλύτερο ποσοστό θα ε, ανακτηθεί το 2011. Να σας πω τρία στοιχεία τώρα που είναι σημαντικά. Για συμβάσεις της Γενικής Διευθύνσεως Έρευνας και Καινοτομίας τέλος το 2008 είχαμε ανακτήσει το 30% των εκκρεμών ποσών αυτό αυξήθηκε στο 55% το 2009 και έφτασε το 68,5% εν έτη 2010. Οπότε η καμπύλη ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση και αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα. Και είναι σημαντικό για μας, πολύ σημαντικό μάλλον εσείς να κατανοήσετε ότι εκεί εστιαζόμαστε, να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Στην πρώτη δουλειά μας στο ελεκτικό συνέδριο Κάθε χρόνο όταν συζητούσαμε την έκθεση πάντα οι ανακτήσεις ήταν μεγάλο σημαντικό ζήτημα για τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου. Όσον αφορά την απλούστευση, ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα, ίσως το θέμα που αντιμετώπισα από όταν έγινε επίτροπος και από ερευνητικού οργανισμούς και από επιστήμονες μεμονωμένους και ερευνητές και επιχειρήσεις είναι το θέμα της απλούστευσης. Όλοι λένε ότι το ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο συνεπάγεται γραφειοκρατία, περιπλοκή και δίκηση. Επιπλοκή και δίκηση. Και γι' αυτό πολλά ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείε κατά τη διάρκεια των καλών οικονομικών καιρών συνειδητά δεν υπέβαλαν αίτηση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα πλαίσιο λόγω όλων των επιπλοκών. Αυτό είναι άκρος θλιβερή απόφαση, ετοιμιγορία όσον αφορά τη γραφειοκρατία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι πρέπει να αντιμετωπίσω. Και το αναγνωρίσατε και στις παρεμβάσεις σας ότι τα πρακτικά βήματα που κάναμε γίνανε όπως αυτά που είπαμε και χτες. Απλοποίηση λοιπόν για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Να πω καταρχάς η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού δεν είναι πλέον θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά δικό σας το Κοινοβουλίου θέμα είναι και το Συμβουλίου. Αυτό θα επιφέρει σημαντικότατη απλούστευση και θα να τη διεξαγωγή σύντομα αυτής της συζητήσεως και να βρεθεί γρήγορα μια λύση. Για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο να σας δώσω μια γεύση των όσων αποφασίσαμε. Πρώτα απ' όλα να δημιουργήσουμε μια, ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την χρηματοδότηση της έρευνας και της ανοτομίας με μια ενιαία ομάδα διαδικασιών συστημάτων πληροφορική κανόνων ανεξάρτητα από το σύστημα χρηματοδοτήσεω. Άρα απλοποίηση της περίπλοκου, του περίπλοκου δικτύου των ποσοστών χρηματοδότησης και του τρόπου υπολογισμού των εμέσων δαπανών. γενικότερη αποδοχή των συστημάτων ε, λογιστικών υπολογισμών των συμμετεχόντων και μέσος όρος του κόστους του προσωπικού. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό που αναφέρατε κατά αποκοπήν ποσά, όποτε αυτό είναι δυνατόν. Η χρηματοδότηση βασίζεται στα αποτελέσματα. Η επιστημονική κοινότητα το βλέπει με πολύ κριτικό μάτι και δεν παρέχει τις λύσεις για όλα τα προβλήματα και απαντήσει σε όλε τι ερωτήσει, πρέπει να διερευνήσουμε κατά πόσε συγκεκριμένε περιορισμένε περιπτώσει θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την προσέγγιση, όπω για τα μικρά προγράμματα. Για ποιο λόγο είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθορίσει κανεί εκ των προτέρων το ακριβέ κόστο που συνεπάγεται ένα ερευνητικό πρόγραμμα και να αποτιμήσει κατά πόσο τα αποτελέσματα που θα επιτυγχάνονται έχουν πράγματι επιτευχθεί. Εν κατακλείδη, ένα πολύ σημαντικά βελτιωμένο σύστημα επιστροφής των δαπανών πρέπει να δημιουργηθεί. Το τρίτο. Αναφερθήκατε στο αποδεκτό επίπεδο σφάλματος και από ό,τι καταλαβαίνω είναι επίμαχο θέμα, Συζητείτε έντονο σε αυτή την Επιτροπή. Δεν είναι ορθό να πει κανείς ότι κατά παρελθόν επειδή τώρα λέμε θα επικεντρωθούμε επί των μεγάλων, πολύ μεγάλων προγραμμάτων με πολύ μεγάλο κίνδυνο, δεν είναι σωστό να λέμε ότι τα μελήσαμε αυτό κατά το παρελθόν. Αλλά για να μπορέσουμε να πετύχουμε το 2% θα πρέπει να πάμε στους μικρούς δικαιούχους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα. Πρέπει να πάμε στους μικρούς δικαιούχους και θεωρούμε ότι θα ήταν πολύ πιο ευνοϊκό αν μπορούσαμε να επικεντρώσουμε τις προσπαθίες μας, το προσωπικό μας, τους πόρους μας κυνηγώντα τα πραγματικά μεγάλα προγράμματα και θεωρούμε ότι είναι σημαντικότατο, κυρίως διότι η ερευνητική κοινότητα συνεχώς μας λέει ότι αυτό είναι ιδιαίτερα επαχθές και αποθαρρύνει τους ερευνητές και τον τομέα από το να συμμετάσχουν στα προγράμματα τα ερευνητικά, χρηματοδοτήσεως μάλλον. Πότε να γίνουν οι χορηγίες ένα χρόνο. Μεσω όρο. Σε εθνικό επίπεδο, περίοδοι κάτω από ένα χρόνο πραγματοποιούνται μόνο για χορηγίες που αφορούν ένα ίδρυμα, για πιο περίπλοκα προγράμματα μεγάλης κλίμακας και με μεγάλη συνεργασία ο χρόνος για τη διάθεση των ποσών είναι συγκρίσιμος με το παρόν ε, πρόγραμμα πλαίσιο, παραδείγματο χάρη. Αν αναφερθώ στο κάτω μέρος που γνωρίζετε καλύτερα, το Γερμανικό ε, Συμβούλιο Ερευνών για τα προγράμματα με συνεργασία πολλών χρειάζεται πάνω από ένα χρόνο από υποβολή της πρώτης γενικής προτάσεως μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. Και η συμβάση για το ε, Ινστιτούτο Ερευνάς που αφορά δοκιμές ανθρώπου σε ζώες θα χρειαστεί και δύο χρόνια μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων. Το ε, πρόγραμμα πλαίσιο 7 τι επιτυγχάνει όσον αφορά τον φορολογούμενο, τι απόδοση έχει όσον αφορά την επένδυση. Αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερος, κυρίως τώρα τον καιρό της λιτότητας, όπου τα κράτη-μέλη λαμβάνουν σοβαρότατα μέτρα οικονομικά που έχουν τεράστιες ε, συνέπειες όσον αφορά τους πολίτες τους και το φορολογούμενο. Λοιπόν, τι έχει αποδώσει το πρόγραμμα. Να πάρουμε το μέσο για την χρηματοδότηση της κατανομής του κινδύνου μας. Είπαν ανεκδοτικά ότι παρήγαγε απίθανα αποτελέσματα, πάρα πολύ καλά αποτελέσματα την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μέχρι ότου έχουμε την ενδιάμεση αξιολόγηση δεν είχαμε συγκεκριμένα στοιχεία που χρειαζόταν και τα στοιχεία δείχνουν ότι για κάθε ευρώ που επενδύεται από την Ευρώπη παίρνουμε 40 ευρώ όσον αφορά το φαινόμενο μόχλευσης. Υπέροχο αποτέλεσμα πρέπει να συνεχιστεί και θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Δημιουργεί ευκαιρίες. Περισσότερα αξιοποιούμε το χρόνο μέσω του προγράμματος αριστείας Πρόσφατα για μία ακόμη φορά είχαμε βραβείο Νόμπελ που ξεκίνησε από αυτό το πλαίσιο και βεβαίως κινητικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την ερευνητική κοινότητα και προφανώς αυτό είναι κάτι που επιφέρει τεράστια ωφέλη. Ίσως σε αυτό το στάδιο θα έπρεπε να σταματήσω διότι ξέρω ότι έχετε περιορισμένα χρονικά περιθώρια. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Η κυρία Ιβανόβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε και την Επίτροπο για την παρουσία της εδώ σήμερα. Νομίζω ότι τα καλά νέα τα ακούσαμε από το ελεκτικό συνέδριο για τη μείωση του ποσοστού σφαλμάτων που είναι ενθαρρυντικά. Αλλά και πάλι τα ανακτηθέντα ποσά ε, είναι ανησυχητικά όπως κατά ε, και εσείς και κύριε Επίτροπε και επεσήμανε και ο εισηγητής μας το 2007 και το 2008 είμαστε στο 50, 51% ε, στις ανακτήσεις ποσών, ενώ για το 2009 είμαστε μόνο στο 47% του συνόλου. τα μέτρα τα οποία σκοπεύει να ε, εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ανακτήσει τα ποσά σε μία από τις ε, γραπτές σας δηλώσεις αναφέρεστε στην, ε, στις συνολικές εντολές ανάκτησης και τις διορθώσεις ποσών. Ε, ειδικά για τα καταποκοπήν ποσά, τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε και γιατί μειώνετε το ποσοστό και πέσαμε από το 51% στο 47% το 2009. Αυτά τα οποία μόλις μας είπατε είναι μεν ενθαρρυντικά, αλλά το ποσοστό ανάκτησης Ε, για το 2010 μας είπατε ότι αυξάνεται, αλλά μπορείτε να μας εξηγήσετε τι έγινε το 2009. Και επίσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τι ακριβώς ε, σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσει την πρόσβαση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για το πρόγραμμα πλαίσιο 7 και για τα άλλα προγράμματα. Σκοπεύετε να αναπτύξετε νέα προγράμματα για να βοηθήσετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ευχαριστώ κυρία Γιάλα Σέντερ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ την Επίτροπο για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε και τις απαντήσεις που μας έδωσε στο ερωτηματολόγιο. Ιδίως αυτή τη σύγκριση που κάνουμε ε, και πολύ συχνά χρησιμοποιούμε για το τι ακριβώς γίνεται στα κράτη-μέλη, τι επιδοτήσεις έχουμε, ε, και με τι ποσά ζει ο κόσμος της έρευνα διότι πολύ συχνά ε, ρίχνουμε το βάρος και το φταίξιμο στους χρόνους χωρίς να κάνουμε σύγκριση μεταξύ αυτών που γίνονται στα κράτη-μέλη όπου εκεί η ερευνητική κοινότητα πρέπει να αντιμετωπίσει και τα περίπλοκα προβλήματα ε, που υπάρχουν στον οικονομικό και χρηματοδοτικό κόσμο και τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να λάβει επιδότηση για τις έρευνές της. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής η σύγκριση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή μεταξύ των ερευνητικών κέντρων που διαχειρίζονται τις επιδοτήσεις ε, με τα χρονοδιαγράμματα τα οποία μας αναφέρεται ένα-δύο χρόνια από τη στιγμή που παρουσιάζεται μία αίτηση μέχρι να ληφθεί υπόψη κτλ. Διαπιστώσατε ότι υπάρχουν διαφορές ή ενδιαφέρουσες καλές πρακτικές ε, που θα μπορέσετε να προσαρμόσετε στους μηχανισμούς χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον κόσμο της έρευνας. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια και εγώ θα ήθελα να φτάσει μια στιγμή στην οποία ε, σε θέματα ανάπτυξης και συνεργασίας η τεχνογνωσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αναγνωριστεί ως κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο. Η δυνατότητα λοιπόν να έχουμε συστήματα ελέγχου και διαχείρισης και αποτελεσματικής χρηματοδότησης ενός πολύ περίπλοκου προγράμματος όπως είναι το πρόγραμμα πλαίσιο θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο οργανωμένο τρόπο τεχνογνωσίας σαν αυτό που θα είχαμε. Αυτή είναι η πρώτη μας τοποθέτηση. και θα ήθελα να διευκρινίσω και το εξής. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε καλά ποσοστά ανάκτηση, διότι δεν υπήρχε σύστημα ανάκτησης. Ήμασταν ικανοποιημένοι γιατί δεν υπήρχε κανένας τρόπος να διαπιστώσουμε εάν υπήρχε κάποιος τρόπος να ανακτήσουμε τα ποσά. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει πλέον ένα σύστημα το οποίο αν κατάλαβα καλά, λειτουργεί, υπάρχουν ανακτήσεις, γι' αυτό και αυξήθηκε το ποσοστό ανάκτηση. Είναι ένα σύστημα επιφυλακής ε, για την ανάγκη να δαπανούμε καλύτερα τα κονδύλια μας. Αλλά, αν κατάλαβα καλά, θεωρούμε ότι ε, μπορούμε να έχουμε και συστήματα μέσω των οποίων μπορούμε να ανακτήσουμε ποσά που στο παρελθόν θεωρούσαμε χαμένα. Ισχύει κάτι τέτοιο. Θα μπορούσαμε να δώσουμε αυτό το καλό νέο και να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλέον συστήματα για τις περιπτώσεις της έρευνας όπου μπορούμε να ανακτήσουμε τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων ε, όταν διαπιστώνουμε ότι δεν έγινε καλή διαχείριση ή ε, εσφαλμένα δόθηκαν κάποια ποσά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, Για το χρόνο τη ε, χορηγίας, το ερώτημά μου ε, καλύφθηκε από την Επίτροπο. Ο κύριος Οντή, λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την υποστημονική κοινότητα και την ερευνητική κοινότητα που είναι η καλύτερη στον κόσμο. Και παραλίγο υπάρξει μεγάλη παρεξήγηση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώσεω και ερευνητών. Και θα ήθελα κυρία Επίτροπε σήμερα να σα ευχαριστήσω Θυμάμαι στην ακρόασή σας δεν είχατε ακόμα αναλάβει τα καθήκοντά σας, δώσατε μια υπόσχεση περί απλουστεύσεως, διότι μας, δώσετε, μας καλέσετε να κάνουμε κάτι σε αυτό το θέμα και δώσατε την υπόσχεση. Είσαστε, κάνετε αυτό που λέτε, το υπόσχεστε, έχετε αυτή την πολιτική προσωπικότητα. Σας ευχαριστώ για αυτό που κάνατε σε αυτή την απλούστευση. Για το ανεκτό επίπεδο σφαλμάτων, ποσοστό σφαλμάτων. Μιλήσαμε το, για το θέμα αυτό το πρωί Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει διάκριση διάκρισης μεταξύ του ανεκτού ποσοστού σφάλματος, που είναι μια έννοια διαχειριστική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια των ευθυνών που έχει για διαχείριση. Από το δεδομένο ελέγχου που αποτελεί για το ελεκτικό συνέδριο. Αυτά τα κριτήρια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και πώς ερμηνεύονται, διότι δεν υπάρχει η ίδια ερμηνεία στα αγγλικά. Χρειάζεται μεγάλη ακρίβεια. Και για το ανεκτό επίπεδο κινδύνου γίνονται συζητήσεις. Χρειάζεται περισσότερος διάλογος. Χρειάζεται λύση. Και για το μέλλον. Και για το παρελθόν. Και κλειπαρώ και εσάς και τις υπηρεσίες και αυτό. Το παρελθόν οδήγησε παρεξηγήσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώσεω και ερευνητική και επιστημονική κοινότητα. Εξού και τρίτη παρατήρηση. Θα συζητήσουμε τι επόμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ. Πώ αισθάνεστε, πώ βλέπετε σήμερα, πού βρίσκονται τα κράτη-μέλη, πού τοποθετούνται όσον αφορά τι συζητήσει περί απαλλαγή, αλλά και περαιτέρω εξευρωπαϊσμού τη έρευνά μα. Σήμερα τα κράτη-μέλη έχουν ανησυχίες, προβλήματα οικονομικά. Πώς μπορούν τα κράτη-μέλη και εμείς να κοινοτικοποιήσουμε κάποιες δημόσιες προσεγγίσεις, όπως η έρευνα. Πώς το βλέπετε. Ξαναεπαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω εκ νέου το ερώτημά μου. να δώσουμε ευρωπαϊκή χρειά περισσότερη στην έρευνά μας. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Όλα αυτά τα περί ανεκτού κινδύνου, Πρόεδρε, είναι περιττές κουβέντες, γιατί δεν υπάρχει αντίληψη για το ποιος είναι ο δικαιούχος. Καλό θα είναι να ξέρει η Επιτροπή πρώτα απ' όλα ποιο είναι δικαιούχο και ποιος ανήκει αυτήν την κατηγορία. Δεν είναι γνωστό λοιπόν αυτό, δεν υπάρχει σαφής ορισμός και γι' αυτό παραμένει και γραφειοκρατική όλη αυτή η δομή και νομίζω η Επιτροπή ότι με αυτόν τον τρόπο έχει και ένα περιθώριο αξιολόγησης μεγαλύτερο. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο εμείς τουλάχιστον έχουμε δείξει μια ευνοϊκή στάση απέναντι στην Επιτροπή, γιατί αν επιμέναμε και, μειώναμε στο 3%, τότε θα έπρεπε στο 5% να ε, εγκατελείπτεται ολόκληρη προσπάθεια και αυτό σημαίνει ότι με το, στο 5% έχουμε μπει ήδη στην, ε, στην κόκκινη ζώνη. Παραμένουμε με το 2-3% στην πράσινη ή γκρίζα. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να πω ότι είμαι ατυχής εισηγήτρια, ατυχής υπογραμμίζω, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα πεδίο στο οποίο σημειώνονται αρκετά προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται, δεν υπάρχουν επαρκείς κανόνες για την έρευνα. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά πάντως πρέπει να πω ότι αυτά τα οποία μας έχει εξασφαλίσει ως δυνατότητες η έρευνα, αυτά που έχουμε μπορέσει να αξιολογήσουμε χάρη στην έρευνα, το streamlining που έχουμε εξασφαλίσει, μας δείχνει ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί κανόνες, αντιφατικοί μερικές φορές και μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να χρειάζεται πλέον να θεσπιστεί ένας γενικός κανόνας ο οποίος θα θέσει εκτός λειτουργίας τους μερικούς ειδικότερους κανόνες γιατί πια δεν έχει, είναι όλοι μεταξύ τους αντικρουόμενοι και δεν έχουν φέρουν κανένα αποτέλεσμα και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μας πει η Επιτροπή τι γνώμη έχει για όλα αυτά και αν σκοπεύει να συνεργαστεί σε αυτήν την υπόθεση. Η κυρία Επίτροπος. Mm. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω με τη σειρά στις ερωτήσεις. Στην ανάκτηση καταρχάς, τι μέτρα σκοπεύουμε να λάβουμε. Στην προηγούμενη επιτροπή, το Δεκέμβριο του 2009, είχαμε μια ανακοίνωση είχε εισαγάγει μια σειρά μέτρων δηλαδή για ουσιαστική απλούστευση και βελτίωση των ανακτήσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρίως με προβολή ε, των ελεγχθησών σε σχέση με τις μη ελεγχθήσεις ε, συναλλαγές ή πληρωμές για τον ίδιο δικαιούχο. Τώρα βέβαια μπορεί ένας δικαιούχος να επιλέξει να, ε, ε, την επιβολή ενός ποσού διορθώσεως κατά αποκοπή σε σχέση με τις ε, κατά περίπτωση διορθώσεις. Και πολλοί το προτιμούν. Εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε να βρούμε μια λύση για μια συνολική διαδικασία ανάκτησης των επιμέρους ποσών μέσα σε μία διαδικασία ανάκτηση, με προστευμένη στο δυνατόν διαδικασία για την Επιτροπή αλλά και για το δικαιούχο. Μικρομεσαίε επιχειρήσει, τι κάνουμε για τι μικρομεσαίε. Κοιτάξτε, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι τεράστια προτεραιότητα, τεράστια προγράμματα προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γιατί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά τη ευρωπαϊκή οικονομία και γιατί είναι εκείνε οι οποίε ε, διαμαρτύρονται περισσότερο για την απουσία απλούστευση. Και με όσα κάνουμε εν γέννη για την απλούστευση, πάλι πρέπει να κάνουμε μερικά πράγματα υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που στην πραγματικότητα να τι προσελκύσουν σε ένα πρόγραμμα ερευνητικό. Με το 15% Φερρυπίν που ακόμη δεν έχουμε επιτύχει αν και πλησιάζουμε. Ε, μπορούμε ιδιαίτερε προκηρύξει σε περιοχέ, ε, τομεί που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προσφέρουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και συχνά το τι σημαίνει αυτό. Μα επιτρέπουν ε, να ορίζουμε κάποιου κανόνε που θα ε, στηρίζουν τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, θα τι προσελκύουν και πάλι σε ένα πρόγραμμα που ενδεχομένω έχουν εγκαταλείψει ή νέε επιχειρήσει και νέου ερευνητέ για πρώτη φορά. Εν πάση περιπτώσει όμω, αν θέλουμε περισσότερη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ερευνητικά προγράμματα, θα πρέπει να απλουστεύσουμε. Και αυτό το επισήμεναν πιστεύω και όλοι οι βουλευτέ τη Επιτροπής σας που έλαβαν το λόγο. Από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο έχω διαπιστώσει εγώ ότι το πιο περίπλοκο πράγμα, η πιο περίπλοκη δουλειά στην Επιτροπή είναι η απλούστευση κύριος ε, Στάις χώρα δεν ακούγεται. Ε, τα έχουμε συζητήσει εδώ και καιρό και ο προκατοχό μου, ο Πίτροπος Ποτότσινικ, είχε κάνει πολλέ προσπάθειε για να ε, εισαγάγει διάφορα στοιχεία πλουστευση στον τρόπο εργασία μας. Είναι ο τομέα ο οποίο έχει λάβει πλέον την κύρια προτεραιότητα, πολιτική προτεραιότητα σε επίπεδο επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 4 Φεβρουαρίου επίση, ε, πρόκειται να συζητήσει το θέμα αυτό με τον πρόεδρό σα, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Μπουζέκ. επίση παρόντα. Και από ό,τι γνωρίζω, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα για το, θέμα αυτό, για την απλούστευση. Επίσης, επίσης ε, απλούστευση σημαίνει και συνέπεια σε όλε τι υπηρεσίε επιτροπέ. Τι σημαίνει αυτό, ότι δηλαδή όταν ένα δικαιούχο έχει να κάνει διαφορετικέ γενικέ διευθύνσει, είναι σημαντικό να αντιμετωπίζεται με συνέπεια και ω προ την προσφορά ε, την ε, υποβολή δηλαδή του προγράμματος, την τελική υποβολή, αλλά και τη διαχείριση μετά το πέρας αυτού. Ο Γενικός μου Γραμματέας λοιπόν εργάζεται σε στενή συνεργασία με τους λοιπούς γενικούς γραμματείς που έχουν στην αρμοδιότητα στα θέματα αυτά, ώστε να εξασφαλίσει συνέπεια στο προϊόν. Αυτό πιστεύω θα θεωρηθεί ευπρόσδεκτο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους λοιπούς εμπλεκόμενους για, τον, ε, για το αποδεκτό ποσοστό κινδύνου. Ε, ο Επίτροπο Σεμέτα, βέβαια, έχει την άμεση αρμοδιότητα στην υπόθεση αυτή. Ξέρω ότι είναι ιδιαίτερα ευγνώμων για τη συνεργασία μαζί σα για τον προσδιορισμό του αποδεκτού επίπεδου κινδύνου, που είναι βεβαίω απαραίτητο και για του ερευνητέ μα όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι έχουν παρισφρήσει κάποιε παρερμηνίε στην υπόθεση αυτή και συνεργαζόμαστε εμεί, ε, η δική μα υπηρεσία, στενά με τι υπηρεσίε του κ. Σεμέτα για να διασκεδάσουμε αυτέ τι ε, παρερμηνίε και βέβαια περιμένουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα και να πείσουμε και εσά στο εγγύ μέλλον για την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων. Επίση, υπήρξε κάποια ερώτηση για το κατά πόσο τα κράτη-μέλη θέλουν ε, με, σε έναν βαθμό να συνδυάσουν του εθνικού ερευνητικού προπολογισμού με τα όσα πράττει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίω, είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, ο ευρωπαϊκό χώρο έρευνα να ολοκληρωθεί και να είναι σε πλήρη λειτουργία στο 2014 τεράστια σημασία σε αυτό, διότι είναι τεράστιος ε, ο κατακαιρματισμός, η επικάλυψη έργου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα ωστόσο να υπογραμμίσω το εξή, ότι αν στραφούμε και κοιτάξουμε τα κράτη-μέλη, τα οποία με πολύ αυστηρές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις αυτή τη στιγμή και περικοπές, ουσιαστικέ περικοπές των προπολογισμών τους, προσπαθούν να κάνουν οικονομίες θα έλεγα ότι αυτά τα κράτη-μέλη, θα επεσήμανα μάλλον ότι αυτά τα κράτη-μέλη είτε διατήρησαν την χρηματοδότηση στην έρευνα, είτε ορισμένα μάλιστα την ενίσχυσαν τη χρηματοδότηση στον τομέα της έρευνας. Μεγάλα κράτη-μέλη όπως η Γερμανία και η Γαλλία δείχνουν και στους τελευταίους προπολογισμού πολύ σημαντικές αυξήσεις στην έρευνα και θα σας παρουσιάσω ως παράδειγμα τη Φιλανδία που ξέρω ότι πολλοί γνωρίζουν αρκετά καλά από τα μέλη της Επιτροπής σας. Στη δεκαετία του 1990 που αντιμετώπισε δεινή οικονομική κατάσταση η χώρα, η κυβέρνηση αναγνώρισε ότι η έρευνα ήταν ένας χώρος που μπορούσε και θέση εργασίας και ανάπτυξη με χάρη στην καινοτομία να προσφέρει και αποφάσισε όχι μόνο να διατηρήσει αλλά και να ενισχύσει τη χρηματοδότηση στην έρευνα. Αυτά τα λέγω πάντοτε όταν συναντιούμε, συναντιούμε με τους ε, υπουργού έρευνα σε επίπεδο Συμβουλίου. Αλλά και από την εμπειρία μου ως υπουργό γνωρίζω ότι εάν δεν αποφασίσει ένας υπουργό με το επιτελείο του, αλλά κυρίως ο υπουργό ως πρόσωπο, ότι είναι κέρια σημασία η έρευνα, εάν δεν δώσει αυτή την προτεραιότητα και πάνω απ' όλα, αν δεν αναγνωριστεί η σημασία και από τα λοιπά Υπουργεία για να δώσω την αντίστοιχη όθηση, δεν μπορεί να έχει την ε, υποστήριξη που χρειάζεται. Και γι' αυτό ελπίζω και στο Συμβούλιο των Υπουργών 4 Φεβρουαρίου ότι θα μπορέσει να δοθεί ένα σαφέ μήνυμα και ε, να αποσταλεί ένα ηχηρό μήνυμα προ του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων για την έρευνα. Ότι η έρευνα δεν είναι δηλαδή μόνο ένα μικρό τομέα ε, πολιτική, δεν είναι μόνο ε, μια προσπάθεια για καινοτομία. Είναι μια οικονομική δραστηριότητα και πολιτική. Και σε μια στιγμή δεινών οικονομικών συνθήκων και αυστηρής λιτότητας θα μπορούμε νομίζω να δώσουμε ένα μήνυμα στους ε, πολίτες ενώ ε, γιατί ενώ σφίγγουμε τα λουριά και τα σφίγγουμε πολύ, υπάρχει και φως στην άκρη του τούνελ. Του αφήνουμε δηλαδή ανοιχτή την άκρη του τουνέλ για να δούνε το φως και να κατευθυνθούν προς τα, προς τα εκεί. Αυτά όπως είπα σε περιόδους δονών οικονομικών ε, προβλημάτων. Επίσης είπα κατά την ε, ομιλία μου ότι ενθαρρύνω όλες τις πλευρές ε, σε συνεργασία και όπως αναγνώρισε η κυρία Γκρέσλη πιστεύω ότι η συνεργασία μπορεί να προσφέρει η συνεργασία και με τις εθνικές αρχές μπορεί να προσφέρει την απλούστευση που χρειαζόμαστε, αλλά εφόσον και οι εθνικές αρχές απλουστεύσουν τις ιστορικές τους διατάξεις. Ε, και για να προχωρήσω θα ήθελα να πω ότι λυπούμε που δόθηκε τέτοια εντύπωση αλλά σας διαβεβαιώ ότι το μόνο που μας, δεν μας διακρίνει είναι απουσία φιλοδοξίας γιατί εμείς θελήσαμε να καταστεί αυτό το έργο η ναυαρχίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο μέσα στην Επιτροπή αλλά και στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αυτή την ε, υψηλή φιλοδοξία και το υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας θέλω να το προαγάγω. Λυπάμαι που δεν είναι ορατό πάντως. Ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να παραμείνουν κύρια προτεραιότητα, ο στόχος του 15% θα επιτευχθεί και πιστεύω ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα ώστε να βεβαιωνόμαστε πώς θα επανέλθουν, θα ενθαρρυνθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ξαναβούν στο πρόγραμμα πλαίσιο. Νομίζω ότι έχω απαντήσει ερωτήσεις στην πλειονότητά τους και φαντάζομαι ότι δεν θα θέλετε να μακρηγορήσω. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θέλω να επισημάνω ότι το πρόγραμμα Euro με επιτυχία. Θα θέλαμε να το συνεχίσουμε και να το αναπτύξουμε. Επίσης πιστεύω, γιατί ήμουν παρούσα στην ε, τελετή των ε, βραβείων Νόμπελ, όπου ένας βραβευθής από το πρόγραμμα πλαίσιο βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ ε, πρέπει να πω όμως ότι βρέθηκα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, σε μεγάλη μηχανία όταν ο καθηγητής ε, έλαβε το λόγο για να ε, καταφερθεί εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέγοντας ότι είναι υπερβολικά γραφειοκρατική βραδεία, δεν αναγνωρίζει το δυναμικό των ερευνητών κτλ. Και ελπίζω να μην ξαναβρεθώ ποτέ σε αυτή τη θέση και να μπορέσουμε να προσελκύσουμε όσο δυνατόν καλούς και ε, δημιουργικούς ερευνητές. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλός ο στόχος αυτός κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ. Κοιτάω πως ε, απευθύνω προς εκείνους που υπέβαλαν ερωτήσεις, είστε ικανοποιημένοι όλοι από τις απαντήσεις που πήρατε. Σας κοιτάω στα μάτια να δω, είστε χαρούμενοι από τις απαντήσεις. Είναι ακόμα εδώ η Επίτροπος, οπότε μπορούμε να τις θέσουμε μια-δυο ερωτήσεις, Σίγκεμπορ. Καλές οι πολιτικές ομιλίες, αλλά <laughs> να έχουν και κάποια ουσία, κυρία Επίτροπε. Κυρία Επίτροπε, το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πολλούς, υπερβολικά πολλούς κανόνες διαφορετικούς. δεν είναι τόσο οι κανόνε για τη συμμετοχή, αλλά ότι είναι αντιφατικοί οι κανόνε μεταξύ των κανόνων συμμετοχή, των δημοσιονομικών κανόνων, των ε, υφισταμένων κανόνων, των δευτερευόντων κανόνων, του τρόπου απόδοση. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα πρόβλημα. Και σε αυτά δεν έχετε λύσει κανένα πρόβλημα των αντίων και πάλι βλέπουμε ότι στηρίζεται τα συστήματα μετά το 2014, πρόγραμμα πλαίσιο δηλαδή, και όλους τους άλλους τομεακούς κανονισμούς με τους ίδιους κανόνες. Τους ξαναβλέπουμε αυτούς τους κανόνες οι οποίοι πάλι είναι σε αντίφαση με αυτά τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε δημοσιονομικά. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Και όσο δεν έχει ρυθμιστεί αυτό, δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει τίποτε. Τέλειωσε. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα όλοι αυτοί οι διαφορετικοί κανόνες, οι κώδικες, τα βιβλία με την νομοθεσία που πρέπει κανεί να λάβει υπόψη του. Θα πρέπει λοιπόν να έχει κανείς ε, ω το δυνατόν πιο απλή εικόνα της κατάσταση και του νομοθετικού πλαισίου. Είναι ε, στον τομέα της έρευνας διαφορετικές οι περιπλοκές, ίσως ναι, αλλά είναι περιπλοκές οι ε, διατάξεις και γι' αυτό δεν βλέπω γιατί μπορείτε να μιλάτε για αποδεκτό ποσοστό σφάλματος. Πώς λέτε λοιπόν ότι όλα είναι ωραία και πρέπει να παραμείνουν ως έχουν. Πρόεδρος. Νομίζω, λέει ο Πρόεδρος, ίσως οι δύο κυρίες θα έπρεπε να βγουν έξω και να το συζητήσουν το θέμα. Ακούστηκε και κάποιο πολιτικό σχόλιο. Θα δώσω το λόγο στον συγγητή. Ε, Εγώ διαφοροποιούμε λίγο προς τις απόψεις μου. Θέλω να πω ότι παρακολουθώ με ενθουσιασμό το πάθος με το οποίο κάνετε τη δουλειά σας, το ότι θέλετε να αλλάξετε τη δουλειά, τα πράγματα, το βλέπω αυτό, Ingeborg. Στον τομέα της έρευνας θέλετε να αλλάξετε μαζικά τα πράγματα. Χαίρομαι. Και χαίρομαι που η επίτροπο και ω πρώην μέλο του Ελεκτικού Συνεδρίου είναι τώρα σε θέση να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα το ζήτημα αυτό. Και το Κοινοβούλιο έχει κάνει σοβαρά βήματα προετοιμασία. Έχουμε την έκθεση Καρβάλιο πρώην ε, ε, Υπουργό, κυρία Καρβάλιο, μάλιστα μέλος τη σα τη πολιτικής ομάδα. Ναι, ναι, διαδέχεται, διαδέχεται. Η, η κυρία Γκρέσλε δεν ακούγεται δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι από τη Βάδη Βιτεμβέργη και κυρίω όχι από τη Βιτεμβέργη, από την οποία κατάγεται η ίδια Ιγκεμπορκ. Εν πάση περιπτώσει, εκεί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σκληρά. Αλλά ε, τέλο πάντων, δυστυχώ δεν ξέρουν τι σημαίνει αισιοδοξία. Παραμένουν πάντα απεσιόδοξοι. Εγώ από, την, ε, από το Σάρλαντ, από τη Σάρλανδη, πάντα αισιόδοξο, πάντα με τη χαρά στα μάτια και βλέπω ότι μπορείτε να προχωρήσετε με επιτυχία. Καλή λοιπόν η παρατήρηση ω προς το Risk Assessment Facility Σα διαβεβαιώ δε ότι εφόσον όλα αυτά τα θετικά πράγματα, αυτή η δυνατότητα της διάδοσης που αναφερθήκατε με το 15, αν και ίσως παραλίγο να πείτε 40%. Και εδώ επανέρχομαι σε μια συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ε, Επενδύσεων. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι ίσως αυτή η διάδοση που λέγαμε το 15% ίσως να έχει κάποιο νόημα ε, γιατί επαναλαμβάνω δεν είναι αναγκαίο οτιδήποτε αυτή τη στιγμή χρηματοδοτείται με δωρεές αποκλειστικά να παραμείνει στο χώρο της δωρεάς. Μπορεί να μεταφερθεί και στην ε, μορφή του δανείου αυτή η ενίσχυση. Και εδώ αναφέρομαι στην ίδια και ω εκπρόσωπο τη Επιτροπή των Προπολογισμών ότι θα μπορούσαμε τότε να έχουμε σημαντική εξοικονόμηση, 50 δισεκατομμύρια σημασία για την αγορά μέσω των δανείων, εάν μετατραπούν αυτέ τι δωρεέ σε δάνεια. Σημαντική απλούστευση, mega simplification program λέει ο στα αγγλικά και νομίζω ότι θα είχε καλά αποτελέσματα και για τη μεσοπρόθεσμη ε, αναθεώρηση της πολιτικής έρευνας πιστεύω μπορούμε να έχουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Πάντως χαίρομαι διότι η Επίτροπος σήμερα εδώ ε, μας δείχνει ότι θέλει να αλλάξει τρόπο πλεύσης, νοοτροπία. Και ως εκ τούτου αισθάνομαι μεγάλη αισιοδοξία και χαίρομαι για την μελλοντική μας συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Επίτροπος θέλει να απαντήσει εκ νέου. Αν επιθυμεί μπορεί, δεν υποχρεούται. Λοιπόν, λοιπόν κοιτάξτε, στο, στο έκτο πρόγραμμα πλαίσιο είχαμε να κάνουμε 2.200 ελέγχους. Αν θέλουμε να πλησιάσουμε το 2% θα πρέπει να φτάσουμε στις 5.200 ε, ελέγχους. Αυτή είναι η συνέπεια λοιπόν η επιπλοκή γραφειοκρατία και το τεράστιο διοικητικό άχθος δεν έφτασαν εν μία ανοιχτή. Κανείς δεν ήθελε να δημιουργηθεί αυτός ο διοικητικός εφιάλτης που έχουμε. Επεξεργαζόμενοι τα διάφορα προγράμματα πλαίσια προσθέσαμε τη χάρπα στα διάφορα πράγματα. Το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πρέπει να μοιραστούμε ε, την ευθύνη. Πρέπει να συνεργαστούν και οι τρει φορεί για να μειωθεί όλο αυτό το διοικητικό άχθος. Λυπούμε αν θεωρήθηκε ότι ήταν πολιτική η ομιλία μου. Δεν είναι. Όπω είπε και ο κ. Χατζημαρκάκης, ε, μιλάω με πάθο γιατί είδα ίδια του τελευταίου μήνε πόσο ε, νευρική, ανήσυχη, απογοητευμένη είναι η επιστημονική και ερευνητική κοινότητα λόγω όλων αυτών. Δεν θα μπω τώρα σε διαφορέ μεταξύ των Ομοσπόνδων Κρατηδίων και το γερμανικό πολιτικό σύστημα. Είναι πιο περίπλοκο από το ίδιο το πρόγραμμα πλαίσιο η πολιτική κατάσταση στη Γερμανία θα αναλάβω την εξή υποχρέωση. Προσβλέπω σε συνεργασία με την Επιτροπή σας προ εξέβρεση λύσεων για να κάνουμε αυτό που είπαν όλα τα μέλη, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, να απλουστεύσουμε τα πράγματα και πιστεύω ότι ο τρόπο στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο είναι ένα σημαντικό μεγάλο βήμα πρόοδου για αυτό το σκοπό. Πιστεύω επίση ότι ο δημοσιονομικό κανονισμό που καθορίζει το πλαίσιο για κοινού κανόνε θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σα ενθαρρύνω λοιπόν να συνεχίσετε με τη δουλειά αυτή και σίγουρα θα έχετε την υποστήριξή μου και συνεργασία μου όπω και το ελεγκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ. Eh, Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Η πρώτη φορά που ήρθατε σε μια ακρόαση σε αυτή την Επιτροπή, τουλάχιστον από τότε που αναλάβατε τη, τα καθήκοντά σας. Σας ξέρουμε όμως από το επαγγελματικό σας παρελθόν, όταν εργαζόσασταν στο ελεκτικό συνέδριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε σήμερα. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η σημερινή μας ημέρα. Φτάσαμε στο τέλος της ακροάσεως των Επιτρόπων. Κύριε Σιγητά, έχετε όλες τις πληροφορίες στη θέση σας. Έχετε μέχρι την 7η Φεβρουαρίου χρόνο για να συντάξετε ένα κείμενο για την έκθεση, ένα σχέδιο εκθέσεω. προσβλέπουμε σε αυτό και μετά είναι θέμα να δημιουργηθούν οι πολιτικέ συμμαχίε. Ελπίζω να μην υπάρχουν εσωτερικέ γερμανικέ διαφορέ, διότι θα πρέπει όλοι να, να αρχίσουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα και θα μπούμε και στι βελγικές διαφορέ και τότε δεν τελειώνουμε άλλο. Ολοκληρώσαμε αυτό το τη της τη διάταξη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ίσως θα μπορούσαμε να διακόψουμε για ένα λεπτό ούτως ώστε η Επίτροπος να μπορέσει να αποχωρήσει και εν συνεχεία προχωράμε στο σημαντικότερο τελικό κομμάτι των εργασιών που έχουμε όσον αφορά το δημοσιονομικό κανονισμό. Eh, να συνεχίσουμε τις εργασίες. E eh, Οι εκπρόσωποι του ΕΛΚ θα μπορούσαν να επαληθεύσουν κατά πόσον ο κύριος Ριβελίνη θα έρθει σήμερα το απόγευμα. Η Ίγκεμπορ Γκρέσλε είναι η συγγήτρια για την Επιτροπή Προπολογισμών. Για την Επιτροπή μας ο εισηγητής είναι ο κύριος Ριβελίνη. Δεδομένου ότι στη συνέχεια έχουμε και συνεδρίαση των συντονιστών, θα ήθελα να ξεκινήσουμε τώρα το κατά πόσο θα έρθει ο κύριος Ριβελίνη. Ε, οψόμεθα, αν έρθει το στο καλύτερο. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από αυτούς που παρακολουθούν τις πολιτικές ομάδες να μας απαληθεύσει τι ακριβώς θα γίνει. Στις 5 και μισή έχουμε προβλέψει των ιστών, αλλά αν τελειώσουμε νωρίτερα θα μπορούσαμε κάλλιστα να ξεκινήσουμε και νωρίτερα τις συνεδρίες των συντονιστών. Αν οι, πολι... οι εκπρόσωποι λοιπόν των πολιτικών ομάδων δουν ότι δεν είναι εδώ συντονιστή τους, ε, ας έρθουν σε επαφή μαζί του ή μαζί της για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε έγκαιρα τη συνεδρία των συντονιστών, γιατί έχουμε χρόνο μέχρι τις 6.30 στη διάθεσή μας. Ίγκεμπορκ, θα ήθελες να κάνεις εσύ μια παρουσίαση για να μα ενημερώσει για το θέμα. Ναι, ευχαριστώ. Είναι σαφή, βέβαια η κατανομή εργασία. Μια μέρα πριν από τις διακοπές, 2010 08, 15 στα γερμανικά σημαίνει μπορεί να είναι οτιδήποτε το επιστητό. Ε, σε σχέση με το recast, δηλαδή την επαναδιατύπωση και την συνθήκη της Λισαβόνας. Ωραίο δωράκι πήραμε για τα Χριστούγεννα. πάση περιπτώσει αυτό έχει προτείνει η Επιτροπή και κράτησε μόλις 7 ε, μήνες ε, το να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει πλέον να ξεκινήσουμε. με αυτή την ε, μορφή του recast. Έχουμε να κάνουμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Έχουμε να κάνουμε περίπου 190 άρθρα του δημοσιονομικού κανονισμού που έχει τροποποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πληθώρα λοιπόν τροποποιήσεων, προτάσεων μάλλον για τροποποίηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πληθώρα νέων διατάξεων που έχουν εισαχθεί. Και Θα θέλω να επισημάνω ιδιαίτερα τα πιο ενδιαφέροντα σημεία όπου η Επιτροπή έχει αναθέσει ουσιαστικά ή σκοπεύει να αναθέσει πολύ μεγάλο κομμάτι αυτών των αρμοδιοτήτων. Η ίδια δεν ξέρω αν έχω καταλάβει τι σκοπεύει να κάνει. τον ιδια δεν ξερω αν εχω καταλαβει απελευθερώνεται για να έχει πιο πολύ χρόνο να δουλεύει. Αυτά. Πολλές επικριτικές παρατηρήσεις. Έχουμε ανάθεση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων της εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού στο σημείο 9, αναφέρεται αυτό. Μετά έχουμε επίσης να κάνουμε για πρώτη φορά με ε, μέσα δημοσιονομικά που όπως είπε πολύ κομψά ο κύριος Χαζημαρκάκης, μας επιτρέπει να εξοικονομήσουμε ένα δις, μπορεί να έρθει μέχρι τα 50 μισή μέσα στις δημοσιονομικέ αγορέ, εφόσον βεβαίω είμαστε σε θέση να αναλάβουμε το σχετικό κίνδυνο. Πράγμα το οποίο σημαίνει βεβαίω ότι, και αυτό είναι αρκετά γελίο, ε, ηρωνικά το, τραγικό, ότι μπορεί να βρεθεί υπόλογος και υπεύθυνο για ε, αποζημίωση ο προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε αποφάσεις στρατηγικές, τις οποίες θα πρέπει να συζητήσουμε πριν ε, καταλήξουμε. Στα άρθρα 23-24 της παλαιάς αρρύθμισης ε, δεν μπορώ να πω τίποτα, έχουν αλλάξει το μεταξύ τα νούμερα τις αποφάσεις για τις οριακέ τιμές τις αναλαμβάνει η Επιτροπή να τις αλλάξει από 15% στο 20%. Στο ανεκτό ποσοστό κινδύνου ή επίπεδο κινδύνου που έχουμε συστήσει αρκετές φορές ε, προβλέπεται ένα μέσον ενημέρωσης και διαχείρισης και προβάλλεται η ιδέα ότι δεν θα πρέπει το Κοινοβούλιο να επιμείνει σε κάποιο ε, όριο θα έπρεπε να είμαστε δηλαδή ανοιχτοί, να βλέπουμε ποιο είναι το όριο σφάλματος και αναλόγως να ζητούμε τις πληροφορίες και τις εξηγήσεις που χρειάζονται. Στο δημοσιονομικό κανονισμό το κύριο άρθρο είναι το λεγόμενο shared management, έμεση δηλαδή διαχείριση. Υπάρχουν πέντε διαφορετικές μορφές διαχείριση μαζί με τις εθνικές οργανώσεις, ε, κοινή διαχείριση το ονομάζεται joint management, indirect management, management, direct management και το καθεξής. Την κοινή διαχείριση την έχει ε, υπαγάγει στην έμεση διαχείριση, indirect management. Και εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια από τα καθήκοντα που έχει ο δικός της ε, Γενικός Διευθυντής ή θα εκχωρούνται στην ε, περίπτωση της κοινή διαχείρισης. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με την περίπτωση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών που συζητήσαμε και που πια δεν έχουν κάνει υποχρέωση λογοδοσία ουσιαστικά άμεσα τουλάχιστον, έχουν όμως έμεσα υποχρέωση λογοδοσίας. αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια πιο συγκεκριμένη πρόταση με τη μορφή ενδεχομένω σύσταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν συζητούμε τις πληροφορίες για την απαλλαγή, τις ε, πληροφορίες τις τροποποίησεις τι οποίε έχει προβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά μας απασχολούν στον τομέα των αρμοδιοτήτων και σε παιδογραμματίες. Αυτό που δεν είναι σαφές είναι το τρόπος χειρισμού του δημοσιονομικού μέσου. Εάν δηλαδή είναι πολύ ασαφές το τωρινό μέσον, οφείλεται στο ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων από τι δραστηριότητε και σε φορολογικού παραδείσους, Φερρυπίν, νησιά και Ιμάν. Και εκεί πέρα ε, γίνονται εμβάσματα που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν. Καλό λοιπόν θα είναι να έχουμε αποφάσεις ε, και πληρωμές οι οποίες θα είναι επιτρεπτές από τους δημοσιονομικούς κανονισμούς και όχι απαράδεκτες και βέβαια ελέγξιμες. Ένα άλλο ζήτημα είναι τα λεγόμενα trust funds, τα καταπιστεύματα που ε, χρηματοδοτούν ε, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την Παγκόσμια Τράπεζα και το καθεξής. Ε, λέμε ότι θέλουμε μέσα στο ψήφισμα για την απαλλαγή να υπάρχουν αυτά τα καταπιστεύματα, να μπορεί να τα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτή τη στιγμή είναι πολύ περιορισμένο το πεδίο δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιορίζεται μόνο σε ανθρωπιστικές δράσεις. Στην εφαρμογή μας του κανονισμού, στο ποιος διαχειρίζεται αυτά τα καταπιστεύματα και ποιος θα πρέπει να συμμετέχει στη διαχείριση, είναι πολύ πιο αυστηρή η διαχείριση στην ίδια διαχείριση, στην απευθεία όπως ονομάζεται διαχείριση των ε, ε, καταπιστευμάτων. Περιμένουμε λοιπόν κάποιε αλλαγέ. Επίση θα έχουμε πολύ άριθμε τροπολογίε από το κομμάτι που αφορά την έρευνα, γιατί πάλι βλέπουμε ότι είναι αντιφατικοί οι κανόνε και θέλουμε να αποφύγουμε αυτέ τι αντιφάσει. Θέλουμε λοιπόν και διατάξει εφαρμογή σαφείς, ορατές, ξεκάθαρες, που θα μπορούν να ενταχθούν στον δημοσιονομικό κανονισμό. Αυτή είναι η κατάσταση προς το παρόν. κάνουμε τις προσπαθίες μας με τις αλλαγές και από τις τελευταίες συζητήσεις που είδαμε και το αποδεκτό, τον αποδεκτό κίνδυνο και την ε, διαχείριση και διαχείριση των μέσων και στην προσοχή συζήτηση που θα συζητήσουμε για τα δημοσιονομικά μέσα και καταμερισμένη διαχείριση κονδυλίων όπου στην καταμερισμένη διαχείριση κονδυλίων έχουμε να κάνουμε με την ανάγκη για ένα ενοποιημένο σύστημα ελέγχου ή μέσων ελέγχου. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει κάνει προκειμένου σημαντικές ε, παρατηρήσεις. Για το κατά πόσο είναι σκόπιμο κάτι τέτοιο. παρατηρήσει που είναι συναφεί και με τόσο είχε πει και η ομάδα εργασία του Συμβουλίου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καλό θα ήταν να γνωρίζουμε ποιο κάνει τι και ποιο φέρει ποια ευθύνη. Πιστοποίηση, θέση πληρωμή, γιατί πρέπει να γνωρίζει κανεί ποιο είναι πιστοποιημένο και υπό ποιου όρου. Και να μπορεί η Επιτροπή βεβαίω να ελέγχει εγκαίρω τι εξελίξει και να μην έρχεται μόνο στο τέλο με μοναδική δυνατότητα παρέμβαση στην την κύρωση του παγώματος των ε, πληρωμών. Αυτά νομίζω πρέπει να συζητήσουμε και με τα κρατημένα, να δούμε και τη δική τους άποψη. Δεν μπορώ να σας πω τίποτε περισσότερο. Ένα μεγάλο εργοτάξιο έχω να σας περιγράψω. Σε βεβαιότητα ότι κάποια στιγμή θα γίνει σπίτι αυτή η έκθεση, αλλά αυτή τη στιγμή η έκθεση μου είναι μόνο ένα εργοτάξιο. Λύθη πλήν θηκέρα μια τάτο ερημένη και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να την έχουμε ε, σε μια σειρά ώστε να δώσουμε συγκεκριμένες ιδέες και ώστε να περιγράψουμε και πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα. Είχαμε 50-60 τροπολογίες ε, υπόψη. Αυτό δεν είναι το ζήτημα ούτε η δυσκολία, αλλά στα μεγάλα θέματα, στα κύρια ζητήματα, πώς διαμορφώνει το έλεγχος, ε, πώς γίνεται ο έλεγχος για την άμεση, για την έμεση ε, διαχείριση, πώς χειριζόμαστε το θέμα των απαλλαγών για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, το ερώτημα του τι κάνουμε, πώς συνεχίζουμε με τα χρηματοδοτικά μέσα, τα καταπιστεύματα, το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου. καλό θα είναι να γνωρίζουμε λίγο περισσότερο ποια είναι η κατάσταση. Δηλαδή τα υπόλοιπα ζητήματα που παραμένουν εκκρέμη είναι μάλλον ασήμαντα ή δευτερεύοντα και μπορούν να επιληθούν. Ευχαριστώ, λέει ο Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία, θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε το άρθρο 51, δηλαδή δύο επιτροπές οι οποίες συζητούν εκ παραλίλου και ψηφίζουν ταυτόχρονα. Ε, η μέθοδος εργασίας λοιπόν ε, ε, είναι ακόμα προς ε, επισημοποίηση. Ο κύριος Χατζημαρκάκης, η κυρία Γιάλα Σέντερ θέλουν το λόγο και μετά να στραφώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι εδώ οι κύριοι Παρίς και Φομπέτερ, δεν ξέρω αν θέλουν να παρέμβουν. Ναι, ωραία. Θα σας δώσω στη συνέχεια το λόγο. Ο κύριος Χατζημαρκάκης, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τη συνάδελφη κυρία Γκρέτσλε, η οποία συνεργάστηκε εντατικά στο μεγάλο αυτό εργοστάσιο με τη συνάδελφο, με τη συνάδελφο Ριβελίνη. Δεν σα λέω, είναι πολύ σκληρή δουλειά που έχει αναλάβει, αλλά είμαι βεβαίω ότι θα την φέρει session πέρα τουλάχιστον εσύ. Το κύριο Ριβελίνη δεν το γνωρίζω τόσο, οπότε ποτέ έρχεται στην ομάδα εργασία, αλλά σπάνια τον έχω δει στην επιτροπή μα. πάση περιπτώσει. Μα δεν είναι Γερμανό, λέει ο Πρόεδρο. Ε, μα γι' αυτό ίσως ναι. Πιο δύσκολα ακόμα. Ιταλό πρέπει να είναι. Ε, πρέπει λοιπόν να δούμε το θέμα και να το συσχετίσουμε με τις δημοσιονομικέ προοπτικές. Μήπω θα πρέπει να γίνει μια στρατηγική συζήτηση εδώ μαζί με την Επιτροπή ε, των Προϋπολογισμών ώστε να δούμε πώ ε, μπορούμε να το συνδυάσουμε με τι δημοσιονομικες προοπτικέ. προοπτικές. Γιατί Ιούνιο-Ιούλιο θα καταθέσει η Επιτροπή της προτάσει για τι δημοσιονομικές προοπτικές και μπορούμε να δούμε ποια είναι τα σημεία αναφοράς, σύμπτωσης ή απόκλησης. Πάντω τα χρηματοδοτικά ε, μέσα έχουν σύμπτώση ή απόκληση. Πάντοτε χρηματοδοτικά μέσα έχουν κεντρική σημασία με προκειμένου το πρωί, η αποκληση παντω τα χρηματοδοτικα μεσα εχουν κεντρικη σημασια εν προκειμενου το πρωι η συζητηση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την έκθεση του κ. Οντή νομίζω έδειξε, έγινε μια ουσιαστική συζήτηση για το πώ θα πρέπει στο μέλλον να χειριστούμε τα θέματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, να της προσδώσουμε μεγαλύτερο έλεγχο, δεν μπορεί βέβαια να, είναι, να εδρεύει στην, ε, στις νήσους Κέιμαν. Και χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει και ένας έλεγχος ουσιαστικός, μια εποπτεία ουσιαστική. Νομίζω ότι βρέθηκε, εξευρέθη μια συμφωνία ή συνένεση καλύτερα για το ποιο θα ήταν το καταλληλότερο μέσον ελέγχου. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε και σε μια διαδικασία απαλλαγή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί χρειάζεται να έχουμε κανόνες ε, οι οποίοι όμω δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα τη δουλειά μα. Αν συγκρίνουμε του κανόνε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία είναι υποχρεωμένη να καταγράφει και τα μαύρα νούμερα, τα μελανά νούμερα δηλαδή, ε, και το πράτη κιόλα, έχει διαφορετική κατάσταση και νομίζω ότι είναι θετικό το ότι έχουμε την ευκαιρία με την κυρία Κλέση να συζητήσουμε όλα αυτά. Έχω πάντως ένα ερώτημα σε σχέση με τον έλεγχο στο άρθρο 75 των απατώμε του τωρινού κανονισμού και θα μας επαληθεύσει και η Επιτροπή αναφέρεται ε, η ανάγκη να συσταθεί ένα ανεξάρτητο ελεγκτικό σώμα. Ποιος, ποιος θα είναι αυτός, ποιος μπορεί να είναι αυτός. Και αν ε, αυτή η φράση εννοεί τους εθνικούς δημοσιονομικούς ελεγκτές, ή κάποιους ιδιώτες στους οποίους προσλαμβάνει, ανεξάρτητος δηλαδή ελεγκτές στους οποίους προσλαμβάνουν οι εθνικές αρχές. Το θέμα είναι πώς θα δρουν αυτοί, θα είναι κατόπιν εντολής του ελεγκτικού συνεδρίου ή ανεξάρτητα τελείω. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε πριν καταλήξουμε σε κάποια απόφαση εδώ. Ίσως θες να πεις δύο λόγια, Ίγκε, αλλά μάλλον η Επιτροπή καλύτερα. Ευχαριστώ κυρία ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Γκρέσλε για τη δουλειά της και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητήσει και με την εισηγήτρια και με τον κύριο Ριβελίνη που φαντάζομαι την επόμενη φορά θα είναι εδώ. Να πιάσω λίγο το νήμα της πρότασης και τα όσα κάνουμε με την κυρία Γκρέσλε και τους συναδέλφους από την Επιτροπή Προϋπολογισμών και να σας πω ότι αυτό το νέο μέσο που έχει και τη θετική διάσταση του γεγονός ότι είναι, το ότι πάρα πολύ ανοιχτό και μας δίνει τη δυνατότητα να αναθεωρήσουμε όλες τις πτυχές οι οποίες ε, είχαμε διαπιστώσει στο παρελθόν ότι χρειάζονταν αναθεώρηση και μας δίνει τη δυνατότητα νομίζω ε, να κάνουμε πράγματα αλλά ταυτόχρονα και τη μεγάλη ευθύνη ώστε να προκύψει το προϊόν που θα πρέπει να προκύψει από την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο και από την κοινή πρόταση των δύο επιτροπών να έχουμε καλύτερη διαχείριση εκ των προτέρων καλύτερη διαχείριση του προπολογισμού και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να κάνουμε και έναν εκ των υστέρων έλεγχο, ο οποίος ε, δεν θα είναι τόσο δαπανηρός ε, ως προς τα συστήματα, αλλά και το προσωπικό των θεσμικών οργάνων που θα το κάνουν. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μία πλούστευση, διότι γνωρίζουμε και μας το λένε και οι τελικοί δικαιούχοι κάθε μέρα ότι τα προβλήματα στη διαχείριση δημιουργούν και ένα μεγαλύτερο κίνδυνο ασφαλμάτων. Δηλαδή τα περισσότερα σφάλματα τα οποία διαπράττονται που δεν έχουν σχέση με την απάτη ή τις παρατυπίες ε, ή την κακυβούληση κάποιων πρόκειται απλώς για λάθη του συστήματος. Επομένως ε, υπάρχει ανάγκη να υπάρχει συνέπεια και συνέπεια όπως έλεγε η κυρία Γκρέσλε προηγουμένως, να ε, έχουμε συντονισμό και με τους υφιστάμενους κανονισμούς. Μιλήσαμε πριν για την έρευνα, αλλά και για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Δηλαδή, για όλους τους κανονισμούς να υπάρχει τουλάχιστον μία απέτηση ε, μια δυναμική που θα πορεύει από τον ε, δημοσιονομικό κανονισμό και θα μας επιτρέπει να έχουμε μεγαλύτερη συνέπεια στις πράξεις μας, αλλά συνέπεια και με τους νόμους των κρατών μελών και με τους κανόνες τους, διότι πολλές φορές οι τελικοί δικαιούχοι μας λένε ότι τα προβλήματα ε, προκύπτουν από το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες κατά την χρηματοδότηση ή τη συγχρηματοδότηση. Υπόκειται δηλαδή σε διαφορετικούς κανονισμούς, σε διαφορετική νομοθεσία, διαφορετικά έντυπα και σε κάποιες περιπτώσεις για τους ελέγχους και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται και υπάρχουν σαφώς και λάθη ε, προς αυτό λόγω αυτού του γεγονότος. Ε, ως προς τον ανεκτό κίνδυνο, νομίζω ότι θα πρέπει να εισαχθούν κάποιοι κανόνες εδώ, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Μπορεί η κυρία Γκρέσλα να αντιμετωπίσει προβλήματα ε, με το σύστημα του σηματοδότη. Ε, το σύστημα του φωτονίου σηματοδότη θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες και στα μέλη του κοινοβολίου ε, να διαπιστώσουν ότι υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος, διότι είναι πολύ πιο εύκολο να το προβάλλουμε και να το εξηγήσουμε. Μία απλούστευση λοιπόν και της επικοινωνίας μας προς, το, προς τα έξω, αλλά και απλούστευση και των διαδικασιών που έχουμε εμείς εκ των έσω. Θα ήθελα επίσης να γνωρίζω διότι εγώ εν μέρη τουλάχιστον συμφωνώ με την αρχική της πρόταση της κυρίας Γκρέσλε και επειδή ούτως ή άλλως ε, Ο πρόεδρός μας ήταν αυτός ο οποίος πρότεινε να έχουμε ένα ευρύτερο όραμα και έχουμε και την τοποθέτηση του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι αλήθεια ότι έχει πιο αυτόνομες θέσεις αλλά λιγότερη αυτονομία ως προς τη ρύθμιση ή τον προπολογισμό όπως συμβαίνει για παράδειγμα με την Ισπανία ή τη Γερμανία. Ε, είμαι υπέρ λοιπόν της αναθεώρησης και να φροντίσουμε ε, σε εθνικό επίπεδο να είμαστε πιο αυστηροί στην εφαρμογή μας. Αποδείχθηκε άλλωστε στην τελευταία απαλλαγή ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που υπογράφουν τη δήλωση αλλά ε, αντιμετωπίζει προβλήματα αφότου γίνεται υπογραφή της ε, εθνικής δήλωσης. Θα πρέπει λοιπόν να είναι χρήσιμο αυτό που έχουμε και θα ήθελα να ακούσω κάποια παραπάνω πράγματα από αυτού. Όσον αφορά τώρα την ε, διαμάχη που υπάρχει μεταξύ των επιδοτήσεων ή των δανείων που θέτει ο κύριος Χατζημαρκάκης, ε, νομίζω ότι θα το έπρεπε, έπρεπε να το εξετάσουμε και αυτό εκ των προτέρων. Ε, δεν νομίζω ότι αργότερα θα γίνει πιο περίπλοκο. Ε, ούτως ή άλλως πρέπει να συζητηθεί με τις τράπεζες και όλη την κατάσταση που είχαμε με τις τράπεζες και το γεγονός ότι τα πράγματα δεν ήταν διάφανα ε, και όλα όσα προέκυψαν για την κοινωνία μας και τα θεσμικά μας όργανα νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ε, όπως είπε και η συγγήτρια επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τη σχέση με την Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων η οποία ε, ε, έρχεται πλέον σε πολύ περισσότερες κοινωτικές πολιτικές και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα με μεγαλύτερη χρηματοδότηση, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να είμαστε συνεπείς ε, και να βλέπουμε και τι γίνεται με τους ελέγχους. Για τους δημόσιους διαγωνισμούς νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ε, απαιτεί περισσότερο ε, προσοχή και μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα και θα έπρεπε ίσως από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε και κριτήρια ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Ως προς το ΦΠΑ και τη συνέπεια νομίζω ότι οι τελικοί δικαιούχοι διαμαρτυρήθηκαν ε, αρκετά συχνά για το τι γίνεται με την επιλεξιμότητα και σε κάποιες περιπτώσεις το ΦΠΑ έχει αλλάξει τελείως τις ισορροπίες της συμμετοχής. Ε, και τέλος το θέμα των υπηρεσιών, το οποίο νομίζω ότι δικαίως η συγγήτρια το θέτει ως προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δει τι γίνεται με το, επίπεδο, ε, με το πακέτο των οργανισμών, ε, σε όλες τις πτυχές ε, για τον πολιτικό έλεγχο. Εγώ από τις μεταφορές έχω πολύ καλά παραδείγματα. Ε, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις οι οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μα ζητά βοήθεια για να ελέγξουμε κάποιους οργανισμούς και δεν είναι οικονομικοί οι λόγοι, είναι πολιτικοί. Θα πρέπει να υπάρχει όμως ένας δημοσιονομικός έλεγχος. Είμαι αδιατεθειμένη λοιπόν να ακούσω τις προτάσεις που μας κάνει η Σύγχυτρη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γιούζο. Eh, ο εισηγητή, ο κύριο Λιβελίνη, κατέφτασε. Λοιπόν, προτείνω να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Οντί και εν συνεχεία ακούμε σας κύριε Λιβελίνη, και μετά επιστρέφουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Οντί. Ευχαριστώ να πω κάτι την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, διότι αναφέρθηκε και παρατείνει την πρωινή μα συζήτηση αυτό. Θα προτείνω μια τροπολογία που ήδη ψηφίστηκε εξάλλου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται μέτοχο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι διακυβερνητικό εργαλείο λοιπόν η, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρειάζεται μεγαλύτερη κοινοτικοποίηση και ένα άλλο στάδιο θα είναι να γίνει τελικά μέτοχο η Ένωση. Ο, πρόεδρο πρόεδρος είναι υπέρ, το Συμβούλιο προφανώ λιγότερο, το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να τοποθετηθεί. Δύο παρατηρήσει όσον αφορά τον κανονισμό. Δεν ξέρω αν είναι καλός τόπος αυτός, δεν είμαι εγώ ειδικό παραπάνω την ίγκε. Στην ίδια λογική των μακροπρόθεσμων επενδύσεων που αντιμετωπίζει η Ήπειρος και ξέρουμε ότι εκφράστηκαν όλων των ειδών οι απόψη επί των επενδύσεων και των λεπτομεριών χρηματοδοτήσεως. Με τα Barroso Bond, τα Juncker Bond, όλα τα ομόλογα, το Project Bond, B, η e iBond κλπ. Μήπως θα μπορούσαμε στην όλη διάθεση του κοινοτικού προπολογισμού στο κεφάλαιο, στον τίτλο 3 κεφάλαιο 2 να θέσουμε ότι υπάρχει ένας τομέας επενδύσεων στις οποίες τοποθετούμε τις μεγάλες πολιτικές παρεμβάσεις όσον όπου έχουν διαφορετική χρηματοδότηση από ό,τι είναι η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεύτερη παρατήρηση αφορά τις προθεσμίες για την απαλλαγή. Ίσως να ακούγεται εν είδη ανεκδότου. Είμαστε Ιανουάριο του 2011 και μιλάμε για λογαριασμό του 2009 και θα ψηφίσουμε μήνα Απρίλιο του 2011. Εγώ θα πρότεινα το εξή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει γνώση της εκθέσεως του λεκτικού συνεδρίου όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Μήνα Ιούνιο του έτους που ακολουθεί το κλείσιμο των λογαριασμών εμείς να ακολουθήσουμε τη διαδικασία μας πολιτικού ελέγχου το δεύτερο εξάμεινο και να μπορούμε να ψηφίσουμε στο Κοινοβούλιο πριν από το έτος που ακολουθεί τον ελεγχόμενο χρόνο. Όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς, τα πράγματα έχουν ξεκαθαριστεί λίγο πολύ. Τι προβλέπετε, τι οι λογαριασμοί θα δίδονται στις 31 Μαρτίου. Θεωρώ ότι είναι βολική αυτή η προθεσμία. Όμως, η υποβολή της εκθέσης του ελεκτικού συνεδρίου προβλέπεται μήνα Νοέμβριο. Πολύ αργά, πολύ αργά. Λοιπόν, μα λένε ότι υπάρχουν προβληματικέ σχέσει με του επιτρόπου, ότι χρειάζεται χρόνο για μετάφραση κλπ. Εγώ θα έλεγα ότι η αποστολή του ελεκτικού συνεδρίου είναι αποστολή μόνιμη. Εγώ δεν βλέπω ποιο πρόβλημα υπάρχει το ελεκτικό συνέδριο να μπορεί αρκετά γρήγορα να εκφράζει κάποιε πρώτε απόψει. Τι θα μάθει τον, από Ιούλιο μέχρι τον Εύετο το ελεκτικό συνέδριο που δεν γνωρίζει τον Ιανουάριο πραγματικά απευθύνω έκκληση τόσο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα διάλογο όσον αφορά αυτές τις προθεσμίες για την απαλλαγή της, τα χρονοδιαγράμματα τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ τραβηγμένα. Κρατούν πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ενδιαφέρουσες ιδέες. Κυρία Ριβελίνη, χαίρομαι που ήρθατε. Κυρία Γκρέσλα έκανε μια βασική εισαγωγή, κάλυψε τα βασικά σημεία Αναφέρθηκε στο όσα κάνετε στην ομάδα εργασία, αυτά που συζητήσατε. Σα δίνω όμω τη δυνατότητα να εκφράσετε τι απόψει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν πρώτη, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, αλλά είμαι εισηγητή για μια γνωμοδότηση στο περιβάλλον για του αρωτές σώματο που ψηφίζουν. Άρα δεν μπορώ ταυτόχρονα να είμαι πανταχού παρόν σε δύο επίτροπε, και μάλιστα μετά πρέπει να πάω να ψηφίσω. Θα με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι, αλλά δυστυχώ ε, ε, γίνονται ταυτόχρονα, εξετάζονται ταυτόχρονα τα δύο αυτά θέματά μου. Πριν να εκφράσω κάποιε σκέψει, επιτρέψτε μου να συμφωνήσω όσον αφορά τι παρατηρήσει του συναδέλφου ΟΝΤΙ, όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα. Διότι ο έλεγχο πιστεύω ότι ο χρόνο του ελέγχου, το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου είναι σημαντικότατο ζήτημα και άκρο επίκαιρο. Όμω επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο νέο δημοσιονομικό κανονισμό και την άμεση και έμεση διαχείριση του προπολογισμού και πιο συγκεκριμένα τα άρθρα 53 και ακόλουθα ε, του νέου κειμένου, του νέου κανονισμού. Τα εν λόγω άρθρα, σαν βασικά χαρακτηριστικά, έχουν την ανάθεση του προϋπολογισμού, το σύστημα του ελέγχου και η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μάλλον Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο και σε σχέση με το παρελθόν διευρύνεται η ανάθεση σε εξωτερικούς φορείς της Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα πιστεύω ότι είναι σημαντικότατο να γίνει ενδελεχής ανάλυση. Πρώτα απ' όλα, θετικές σκέψεις. Κάτι θετικό. Η μείωση του άχθους για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θετική επίσης η μείωση της επιρροής του Κοινοβουλίου επί της αποφάσεως, επί των αποφάσεων, αλλά κυρίως του ελέγχου των πόρων, αλλά επιτρέψτε μου να θεωρήσω κάτι αρνητικό την απόφαση μιας έλλειψης σαφού, σαφούς ορισμός όσον αφορά την αλυσίδα των ευθυνών του ελέγχου. Υπάρχει λοιπόν, εν τη αυτή περιπτώση, ε, μικρότερη διαφάνεια όσον αφορά τα λογιστικά. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι πρώτες Ευρωπαϊκής Επιτροπής σίγουρα οδηγεί σε εξορθολογισμό του διαχειριστικού συστήματος και του ελέγχου του τομέα της γεωργίας. Η πρόταση άλλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταξύ άλλων απλουστεύει και την ορολογία και αυτό είναι σίγουρα θετικό. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαχωρίζεται μεταξύ του οργάνου πληρωμών και του οργάνου πιστοποίησης στη Γεωργία και τα, τα συγχωνεύει και δημιουργεί ένα φορέα. Και ταυτόχρονα δημιουργείται ένα οικοδόμημα ενδιαμέσων φορέων που μπορούν να είναι ενδιάμεση φορείς μεταξύ των διοικητικών φορέων των κρατών μελών. Και προτείνεται η εισαγωγή μιας δήλωσης αξιοπιστίας αλλά όχι εθνικές δηλώσεις. Αυτό προσφέρει βελτίωση της διαχείρισης των ευθυνών, αλλά όχι των φορέων που ακολούθως μπορεί να επιφορτιστούν με τη διαχείριση των πόρων, των ευρωπαϊκών. Τέλος, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι αυτή η πρόταση θεσπίζει νέα άρθρα σε σχέση με τον παλιό κανονισμό. Τα άρθρα 54 και 53 τα εντάσσει και ακυρώνει τρεις ρυθμίσεις διαχείρισης. Στην παρούσα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται η έμεση και η άμεση διαχείριση μόνο. Όσον αφορά την άμεση διαχείριση, πιστεύω ότι οι ρυθμίσεις μοιάζουν πολύ με τις παρελθούσες Τίποτα δεν αλλάζει λοιπόν σε σχέση με τον πρώτερο δημοσιονομικό κανονισμό. Όμως, όσον αφορά την έμεση διαχείριση, ε, έχουμε διάφορες ποικίλε καινοτομίε. Η πιο ενδιαφέρουσα βασική καινοτομία είναι ότι οι δημοσιονομικοί, οι χρηματοσυντητικοί οργανισμοί, οι τράπεζες, οι επενδυτικές τράπεζες, δύνανται να χρησιμοποιήσουν τους πόρους του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για ε, δημοσιονομικά μέσα ε, και για, την και για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και κάποιο που υπενθύμησε την καινοτομία τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που μπορεί να συμμετέχει ε, με νέο τρόπο το Κοινοβούλιο στο... στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Βασικό ερώτημα. Και ελπίζω να μπορεί να το διευκρινίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι το εξή. Αν θέλουμε να διευρύνουμε το εύρος, των, αν θέλουμε να το, τις εξουσίες που έχουν αυτοί οι φορείς. Διότι φαίνεται να δίνουμε πολύ το ελεύθερο σε αυτούς τους φορείς να χειρίζονται το ευρωπαϊκό χρήμα. Όλοι μπορούν να το χειρίζονται, αλλά προσοχή, εκτός όμως των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι το θεμελιώδες σημείο που σήμερα πρέπει να ξεκαθαρίσει και να διευλευκάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο νέο κανονισμό που πρόκειται να εγκρίνουμε, που καλούμε θα να εγκρίνουμε. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Τσέσκοβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που παίρνω το λόγο σήμερα, αλλά ε, παρακολούθησα πάρα πολλά σημεία και θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες για τη συζήτηση. Ε, για αυτά τα νέα χρηματοδοτικά μέσα, διότι πραγματικά μας δίνονται νέα στοιχεία και μπορούμε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντί παρά το γεγονός ότι είμαστε από διαφορετικέ πολιτικές ομάδες, θα πρέπει να σας πω ότι σε γενικέ γραμμές συμφωνώ με τα όσα είπατε. Και θα ήθελα επίσης která se vlastně neustále vrací k... Να κάνω σήμερα μία σειρά από σχόλια για θέματα στα οποία επενερχόμεθα συνεχώς. Παραδείγματο χάρη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το θέμα των ευρωομολόγων. Όπως ε, ακούσαμε σήμερα, με καθησυχάζει το γεγονός ότι εμφανίστηκε αυτή η ιδέα των project bonds. Θεωρώ ότι αυτά τα νέα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία ε, εμφανίζονται θα μπορέσουν να είναι χρήσιμα και σε πολιτικό επίπεδο, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε πώς μπορούμε να ε, προσδώσουμε ένα πιο ευρωπαϊκό χαρακτήρα σε όλα αυτά τα ε, όργανα στα οποία αναφερόμαστε, κυρίως για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ελπίζω η συζήτηση στην Επιτροπή μας να συνεχίσει γιατί είναι ιδιαίτερα επικοδομητική αλλά ε, πραγματικά θεωρώ ότι το θέμα των κρατών μελών σε ατομικό επίπεδο είναι πολύ σημαντικό. Ο ρόλος που έχουν τα κράτη-μέλη τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν ε, κάλεστα να είναι μέτοχοι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στην Ευρωπαϊκή ε, Κεντρική Τράπεζα, ε, σε διάφορα χρηματοπιστωτικά όργανα αυτής της μορφής. ακόμα και η Επιτροπή μας θα μπορούσε να ε, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και να αποτελήσουμε και το κινητήριο μοχλό που θα μπορούσε να δώσει μια νέα όθηση ε, στα όργανα αυτά. Ε, όσον αφορά τώρα τις προθεσμίες, ε, το ανέφεραν και οι συνάδελφοι, καλό θα ήταν να μειωθούν κάποιες προθεσμίες. Παραδείγματος χάρη για την έγκριση ε, μιας διαδικασίας. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι ε, στο παρελθόν, κατά την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, πριν ε, γίνω ευρωβουλευτής, ε, ήμουν λογίστρια ε, και έκανα τέτοιους ελέγχους και μου δόθηκε ευκαιρία και στο παρελθόν να συζητήσω με πολλούς πολιτικούς στην τσεχική δημοκρατία, στη χώρα μου. Και από αυτή την εμπειρία διαπίστωσα ότι πολλές φορές χρησιμοποιούνται ε, χρηματοπιστωτικά μέσα για διάφορα κονδύλια. Πολύ συχνά, δε, όχι μόνο εδώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί μια διαδικασία ελέγχου ε, ακόμα και με ιδιωτικές επιχειρήσεις, ακόμα και με επιχειρήσεις που ορισμένες φορές είναι δικαιούχοι και λαμβάνουν κάποια επιδότηση. Για να ολοκληρωθεί λοιπόν μια διαδικασία, ένα λογιστικό έτος ε, να κλείσει και να γίνει ο έλεγχος, αυτή τη στιγμή έχει περάσει ε, το δημοσιονομικό έτος ε, είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη διότι ε, παρεμβαίνω στο τέλος αυτής της συζήτησης αλλά αν κατάλαβα καλά Ναι, μεν είναι φυσιολογικό να συζητάμε ε, για το 2009 και την απαλλαγή για τα όσα δαπανήθηκαν στο έτος αυτό, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένα περιθώριο να συζητήσουμε τα πράγματα βαθμιδών, να αναλύσουμε σιγά σιγά ε, τα πάντα, να μπορέσουμε να δούμε όλους τους δικαιούχους, όλα τα στάδια, ε, όποιοι και να είναι αυτοί, αν είναι πόλεις, επιχειρήσεις, ε, περιφέρειες, οτιδήποτε θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να ε, εξισορροπήσουμε κάποιος αυτή τη διαδικασία έγκρισης της, ε, του προπολογισμού. Και η εμπειρία που έχω στον ιδιωτικό τομέα ε, αυτό μου λέει. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, αισθάνθηκα κάπως δύσκολα εκεί που ο κύριος Οντί Θεώρησα ότι κάπου μπερδεύτηκε. Α, κατάλαβα όμω, Ξεκαθαρίστηκα τα πράγματα. Κυρία Κρέστλε, εν συντομία και μετά το λόγο θα τον έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήθελα να αναφερθώ πάλι στην ΕΤΕ και κατά εξαίρεση να προστατέψω τη φήμη της Επιτροπής γιατί δεν νομίζω ότι κάνει τόσο κακά τη δουλειά της στην Επιτροπή. Να το πω με αυτό. Μη τι άλλο είναι εδώ, κάθονται, μας ακούνε, κάπως επηρεάζουμε την ΕΤΕ, ούτε τους βλέπουμε, ούτε μας ακούνε. Όλες οι αντιπροσωπείες ασχολούνται ακριβώς με αυτό, με το γεγονός ότι βρίσκονται εκτός του ελέγχου. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ασχολείται ακριβώς με επενδύσεις σε φτωχές χώρες ανά τον κόσμο. και δεν μπορεί να υπαχθεί στον έλεγχο το και πρόκειται να το κάνει. Άλλωστε ούτε τους ε, μισθούς τους μπορούμε να ελέγχουμε ή να παρακολουθούμε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει η ΕΤΕ και τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή. Ούτε 400 άτομα δεν έχουν επιτόπου στα τρίτα κράτη θέλω να πω, έξω από την έδρα τους. Η Επιτροπή έχει χιλιάδες προσωπικό διαφορετικές δυνατότητες ελέγχου, διαφορετικό το επίπεδο της δουλειάς μπορούν να κάνουν. Καθήκον μου λοιπόν είναι εδώ να εξασφαλίσω απόδοση λογαριασμών για το φορολογούμενο, για την Ευρώπη και για τον κόσμο. Και θέλω να αποτρέψω κάθε κίνδυνο για τα ευρωπαϊκά κονδύλια όχι κινδύνους που είναι απίθανοι, όχι υπαρκτούς και ουσιαστικούς κινδύνους, θέλω να τους αποτρέψω στην μην δυναμή τα κονδύλια του Ευρωπαίου φορολογουμένου. Ναι, είμαι κάπως της παλαιάς σχολής. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορεί να έχουν εισπράξει μέχρι και 50 εκατομμύρια. Σε άλλες χώρες θα ήταν ίσω και στη φυλακή τέτοιοι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν καλό θα είναι να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα από τι προκλήσεις αυτέ, αλλά και να αποτρέψουμε κάθε κίνδυνο για, τα, για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, γιατί πρέπει για τελευταίο του ευρωπαϊκού φορολογούμενου. Uh, Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρος. Μακρά η ανταλλαγή απόψεων, πολλά σχόλια ακούστηκαν. Στρέφομαι προ την Ευ... Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο κ. Φον Πίτερ. Θέλετε να μιλήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω πρώτο. Είμαι λογιστή στο θεσμικό όργανο και είμαι υπεύθυνο για τη δικασία τη απαλλαγή. Θα προβώ σε κάποια σχόλια από αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Και μετά ο κύριο Παραντή, που είναι ο διευθυντή επιφορτισμένο με την αναθεώρηση δημοσιονομικού κανονισμού, θα αναλάβει τη σκητάλη. Απαντώντα προ τον κύριο Χατζημαρκάκη για το άρθρο 56. Πολύ καλό το ερώτημά σα. Independent Audit Body, τι σημαίνει αυτό, ανεξάρτητος ελεκτικός φορέας. Εκ προθέσεως παρέμεινε αόριστο αυτό, διότι σε κάποια κράτη-μέλη ε, το ανώτερο ελεκτικό όργανο θέλει να παίξει ρόλο και σε άλλα κράτη-μέλη δεν θέλει. Εάν είναι ελεκτικό συνέδριο, το ανώτατο ελεκτικό όργανο είναι ανεξάρτητο ή δεσμεύεται από κανόνε, από άρθρα του δημοσιονομικού κανονισμού, ήταν το ερώτημα. Σε αυτή την άποψη, ο ανώτατο ελεκτικό φορέα ενό κράτου θα παίξει ένα ρόλο όσον αφορά το γενικό εσωτερικό σύστημα ελέγχου που δημιουργείται το δημοσιονομικό κανονισμό. Θα δρά ω τμήμα του εσωτερικού ελέγχου και του σχετικού συστήματο. Και δεν θα είναι ανεξάρτητο για του σκοπού αυτού του έργου, του συγκεκριμένου αλέος θα παρέμενε βεβαίως, βεβαίως ανεξάρτητο. Αλλά α, θέλει να παίξει ένα ρόλο εντός του πλαισίου του εσωτερικού ελέγχου ε, ελέγχοντας δηλώσεις ε, κλπ για να βοηθήσει τις εθνικές δηλώσεις τι είδου θα είναι η δήλωση δεν ξέρουμε, αν θα είναι διαχειριστική φύση ή πολιτική, το συζητάμε. Αλλά χάνει την ανεξαρτησία του φορέα. Ο εξωτερικό ελεγκτή, εν τη αυτή περιπτώση, είναι μόνο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο κύριο Ντί, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για την απαλλαγή, να σε την προσοχή επί το εξή, ότι 31η Μαρτίου αφορά μόνο του προσωρινού λογαριασμού. Αυτή είναι η διαθέσιμη. Πρέπει να ενοποιήσω όλα τα θεσμικά όργανα και τα bodies που μπαίνουν σε αυτό το πλαίσιο και 31η Μαρτίου ίσα ίσα τα καταφέρνουμε. Αντίθετα, 31 1 Ιουλίου είμαστε πιο άνετα για του τελικού λογαριασμού. Λίγο λέω, ε. Υπογράφω συνήθω πριν στην βελγική εθνική γιορτή, όσο υπάρχει αυτή, εθνική επέτειο, το λέω και στον κύριο Στά. Όπω και εκείνο είναι. Και όπως εγώ, είναι και εκείνο Βέλγο. 11 Ιουλίου είναι η φλαμαδική γιορτή, 15 Λοιπόν, θα πρέπει εκεί, θα είναι πρόκληση να υπογράψουμε. Έχουμε τη γαλλόφωνη εθνική γιορτή που είναι 14 τον Ιούλιο, έχουν πολλές εθνικές γιορτές και παίζει το πράγμα. Λοιπόν, αν για τους λογαριασμούς λοιπόν υπάρχουν ήδη στόχοι, ημερομηνίε σαφείς, με λίγα περιθώρια όσον αφορά τους τελικούς λογαριασμούς, αλλά όχι τους προσωρινούς, αν έχετε την άποψη του ελεκτικού συνεδρίου, φανταστούμε, δεν μιλώ εκ μέρου του ελεκτικού συνεδρίου. Αν υπάρχει νομοδότηση τον Ιούλιο, λαμβάνοντα υπόψη ότι διακόπτει μήνα Αύγουστο το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να εργαστεί πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ για να καταλήξει σε μια απαλλαγή το Δεκέμβρη. Βλέποντα ε, την εσωτερική διαδικασία του Κοινοβουλίου, αυτό θα πρέπει να εξεταστεί εκ του σύνεγγυ πριν κανεί ε, αποπειραθεί να θεσπίσει τέτοιο χρονοδιάγραμμα. Κάθε άλλη σκέψη δεν τίθεται καν. Το Ελεκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχουν κάποιες ωτεραιότητες, αλλά θα πρέπει να προσέξετε τις διαδικασίες εντός του χρονοδιαγράμματος του Κοινοβουλίου. Το Ελεκτικό Συνέδριο υποβάλλει την έκθεση αρχές Νοεμβρίου και ψηφίζεται την απαλλαγή τέλος Απριλίου, τώρα. Θα έπρεπε να βραχυνθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα κατά πολύ αν θέλετε να τηρήσετε, δεν θα έλεγα τις 20 Σεπτεμβρίου που πρότεινε η κυρία, που είναι πολύ φιλόδοξη ημερομηνία, αλλά είναι θέματα τακτικής, τα προνόμια σας ως αρχή της απαλλαγής ε, και, ποια, και, πώς ε, ταιριάζουν με τα προνόμια σας ως δημοσιονομική αρχή. Ο κ. Βενιέ ήταν υπέρ της ευθυγραμμίσεως εν γέννη των ελεκτικών διατάξεων επί εκείνων που ισχύουν για τη Γεωργία. Επιθυμίζω ότι έχουμε επίπεδο ασφάλμα πολύ χαμηλό από τη στρατιωτικά ταμεία, παρόλο που τα ταμεία βεβαίως έκαναν μεγάλη πρόοδο φέτος στη Γεωργία. Δεν θα δώσω στοιχεία, αλλά είμαστε πολύ πιο χαμηλά. Όπως είπε η κυρία Γκρέσλε, που η κυρία Γκρέσλε με συγκλώνησε λίγο. Ε, ε, κοιτάξτε, δεν είναι ότι διαλέγουμε, εργαζόμαστε, επεξεργαζόμαστε το θέμα, εργαζόμαστε πολύ, δεν είναι πάρκο αναψυχής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόθεσή μας είναι να διευκρινίσουμε το ρόλο και τις ευθύνες όσον αφορά την ανάθεση, την εκχώρηση της ε, ανάθεση των ευθυνών είναι θέμα μεγέθου υπολογισμού και μεγέθου υπηρεσιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα το συζητήσουμε και περαιτέρω. Θα συζητήσουμε τι τεχνικέ λεπτομέρειε, θα καταλάβουν τι επιθυμίε σα τότε, πιστεύω. Έχετε θεμητέ επιθυμίε. Κάθε διευκρίνηση τεχνική φύση είναι ευπρόσδεκτη. Θα πρέπει ο καθένα να έχει σαφεί ευθύνε. Θέλουμε βελτιωμένο πλαίσιο. Για την απαλλαγή κυρίω. Θα σταματήσω εδώ και ο Ερικ θα πάρει τη σκητάλη και συνεχίζει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να δώσω κάποιες απαντήσεις καταρχάς στις προκατακτικές παρατηρήσεις της κυρίας Γκρέσλε. Η οποία μας κατηγόρησε πως χρειάστηκαν 7 μήνες για να καταλάβουμε πρέπει να υποβάλλεται κάθε στο δημόσιο σκηνικό. Προσδίρισαμε, με πάση περιπτώσει, την ε, περίοδο της ε, τριετίας. Πολλά άρθρα είδαμε. Αλλά δεν σκοπεύουμε το, να περιορίσουμε το δικαίωμα μεταρρύθμισης. Και ύστερα από μια διεξοδική ανάλυση καταλήγουμε Στην εύτη πρόταση για κανονισμό που συνοψίζει τα όσα προκύπτουν απευθεία από τη Λισαβόνα, τι εφαρμογή δηλαδή τη της Λισαβόνα. Και τα διάφορα άρθρα. καθώς και τις προτάσεις μας. Παρατηρώ με αναποίηση ότι θέλουν οι δύο επιτροπές και ο κύριος Ριβελίνη και η κυρία Γκρέσλε να εργαστούν γρήγορα. Και θα απαντώ στον κύριο Χατσμαρκάκη προς τον συσχετισμό με τις μας ε, νομικές προοπτικές πως είναι σημαντικό για μας να υπάρχει ταχεία, υπάρξει ταχεία συμφωνία μεταξύ μου και του Συμβουλίου και βέβαια και με τη βοήθεια, με τη συνδρομή της Επιτροπής ως προς κανόνες εκτέλεσης του προπολογισμού. Και γιατί, διότι ακριβώς θέλουμε να ε, πλαισιώσουν αυτοί οι κανόνες, του τομεακούς κανόνες που θα εμφανιστούν στα μισά του χρόνου, ιδιαίτερους κανόνες προς την έρευνα, τα διευρωπαϊκά δίκτυα και το καθεξής. Άρα, τον, όσο πιο νωρίς έχουμε συμφωνία για την ε, ε, γενική για, ρύθμιση για το γενικό κανονιστικό πλαίσιο, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις ε, συγχύσεις ή αντιφάσεις με τους ε, τομεακούς κανόνες. Θα ήθελα επίση να σημειώσω ότι πολλοί ήταν οι κανόνε που. πολλά ήταν τα προβλήματα που επεσημάνθηκαν. Θα ήθελα να δώσω κάποιε απαντήσει. Αλλά το σημαντικό νομίζω είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί με του εισηγητέ, όπω άλλωστε έχουμε ήδη πράξει. Στην κυρία Γκρέσλε και τον κύριο Ριβελίνη έχουμε ήδη δώσει το σύνολο των προτάσεων μας. Υπάρχει πάνω από 100 σελίδε με επεξηγήσει, ε, ερωτήματα που και η Επιτροπή Προπολογισμών έχει θέσει και στα οποία δεν θα μπορούσα να δώσω αμέσω απάντηση σήμερα, αλλά πάντω ε, εγγράφονται μέσα στον κανονισμό. Και αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε με την τριετή αυτή αναθεώρηση θα ήταν να απλουστεύσουμε τα πράγματα, δηλαδή να βρούμε κανόνες απλούς, σαφείς, προσανατολισμένους προς το αποτέλεσμα, έτσι ώστε οι δικαιούχοι των Ευρωπαϊκών Ταμείων να βρουν τη θέση τους. και να αποκομίσουν στο δυνατόν περισσότερο όφελος. Άρα λοιπόν απλούστευση κανόνων, ναι. Έγινε πολλής λόγος και για το αποδεκτό ποσοστό σφάλματος, η επίπεδο σφάλματος και εδώ πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ ελέγχου και επιπρόσθετου κόστους που μπορεί να επιφέρει αυτός ο έλεγχος, έτσι ώστε να έχουμε έλεγχο βέβαια αποτελεσματικό προς το κόστος του. Και ένα τρίτο στοιχείο, το οποίο κάποιοι από σας ανέφεραν, η διαφοροποίηση του τρόπου παρέμβασης. Η Επιτροπή ήδη αναθέτει πολλά και υπάρχουν πολλές μορφές εκχώρησης ήδη, ανάθεσης ήδη μια σειρά από μέτρα εποπτείας φυσικά, γιατί η Επιτροπή δεν αναθέτει καθήκοντα εκτελεστικά, εάν δεν είναι βεβαία ότι ο εκδοχέας θα κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Και έτσι, τα δημοσιονομικά μέσα, χωρίς να είναι επιδοτήσεις Ήδη αναφέρονταν στον δημοσιονομικό κανονισμό, τέλο πάντων τώρα είναι χωριστά. Υπάρχει ένα άρθρο 120, αυτο και τελέσχε μοναδικό, 120β στην αναπελαία πρόταση, το οποίο προσδιορίζει ένα γενικό πλαίσιο αυτών των δημοσιονομικών μέσων. Η Επιτροπή εργάζεται πολύ με βάση αυτά, τα δημοσιονομικά μέσα, και είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε ουσιαστικά με τα περιορισμένα δημοσιονομικά μέσα που έχουμε στη θέση μας. Ιδιαίτερος δεδομένων των προθέσεων κάποιων κρατών μελών ε, για τις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές. Και υπάρχει και ένα θέμα το οποίο κρίνει θετικά η κυρία Γκρέσλι για το ευρωπαϊκό καταπίστευμα αντί να μετα φέρουμε ή να αποστείλουμε όλα τα χρήματα σε ένα καταπιστεύμα των ΗΠΑ Προτείνουμε τώρα να θεσπίσουμε ένα καταπιστεύμα ευρωπαϊκό. Και επίση υπάρχει και ένα θέμα με την κοινή διαχείριση, στο οποίο έχουμε συζήτηση επιμακρών με τα κράτη-μέλη, τα οποία θεωρούν ότι είναι επαναστατική, και ρηξικέλευθη εξέλιξη ω προ τα διαφορετικά ταμεία. Εμεί δεν τη θεωρούμε τόσο επαναστατική. Απλώ πιστεύουμε ότι με τι υφιστάμενε τομέ μπορούμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, αυτό το οποίο ζητούμε με τον ε, δημοσιονομικό κανονισμό και νομίζω ότι η κύρια καινοτομία στην ε, κοινή αυτή διαχείριση είναι να ζητούμε από αυτούς που ε, διαχειρίζονται τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να, να τους να προβαίνουν σε μια δήλωση αξιοπιστίας που είναι ένα βασικό στοιχείο πιστεύω όταν έχουμε να κάνουμε με έλεγχο και διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Κάποιε παρατηρήσει έχουμε μου επιτρέπετε τώρα, συμπληρωματικέ. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καταρχά. Βεβαίω θα χρειαστεί καλύτερο έλεγχο. θα χρειαστεί ένα, ένα ειδικό καθεστώς, έχει ειδικό καθεστώς δυνάμει τη συνθήκη. και το να συνεργαστούμε περισσότερο από την ήδη πράττουμε με την ΕΤΡΕ μας φάνηκε καλή ιδέα. Και το Risk Sharing Financing Facility, το μέσο το οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα, ουσιαστικά φέρνει καρπούς, λειτουργεί ικανοποιητικά. Είναι ένα καλό παράδειγμα λοιπόν Πιστεύω ότι μπορούμε να δείξουμε στους ε, συνομιλητές μας, ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε για το δημοσιονομικό κανονισμό, με βάση αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Risk Sharing Financial Facility, ότι μπορούμε να εμπνευστούμε κάτι το δημιουργικό. Και με τις προσεχείς δημοσιονομικές ε, προοπτικές θα προσπαθήσουμε να δούμε εάν υπάρχει δυνατότητα για άλλα μέσα εξίσου αξιόπιστα, μέσα τα οποία θα μας επιτρέψουν ε, να εξασφαλίσουν περισσότερα κονδύλια με τη μορφή του δανείου και όχι της δωρεάς για τους ερευνητές, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οποιονδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις θέλουν να αποδηθούν σε κάποιες πιο επικίνδυνες ε, δραστηριότητες. Αυτά. Δεν ξέρω αν η κυρία Γκρέσλη έχει κάτι άλλο να πει. Θα ήθελα απλώ να σημειώσω για τα δημοσιονομικά μέσα για τα οποία έγινε πολλή λόγο ότι θα προσπαθήσουμε στην πρόταση να συμπεριλάβουμε κάποια μέτρα που θα ε, αποτρέπουν την κατάληξη ή τον προορισμό των ίσων καημάν για τα χρήματα αυτά. και προσδιορίζεται ότι θα πρέπει οτιδήποτε διατάξει ενός αστυνομικού κανονισμού να σέβονται τις διατάξεις ε, σχετικές με την ορθή διαχείριση, την αποτροπή του οργανωμένου εγκλήματος, της νομιμοποίησης της εσόδων κτλ. Είναι μια πρόταση την οποία έχουμε καταβαθέσει. εάν γίνει δεκτή και από την νομοθετική αρχή, θα πρέπει βέβαια και να τηρηθεί. Πράγμα το οποίο βέβαια απαιτεί και διαρκή επιτήρηση και παρακολούθηση. Αυτά σε πρώτη δόση. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με τους ηγητές, να προσπαθήσουμε να τους δώσουμε απαντήσεις το ταχύτερο δυνατό και βέβαια να τους βοηθήσουμε στην έκθεσή τους. Ευχαριστώ πολύ. Ε, στρέφουμε προς το ελεγκτικό συνέδριο τώρα. Είδα ότι παρακολουθήσατε με ιδιαίτερη προσοχή. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε και κάποιες παρατηρήσεις και κατόπιν να ακούσουμε την εισηγήτρια για συμπεράσματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκτός εμού έχουμε και άλλα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου εδώ και θα μιλήσω διότι αναφέρθηκε το ελεγκτικό συνέδριο αρκετές φορές. Πράγματι το ελεγκτικό συνέδριο απέστειλε ένα σημείο, το οποίο σχολίαζε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ισχύει κάτι τέτοιο. Το τελευταίο σχόλιο ή συνεισφορά για μένα ήταν λίγο τραβηγμένο, αν μου επιτρέπετε. Χρηματοδοτικό μέσα και οι άλλες πτυχές οι οποίες συζητήθηκαν δεν αποτέλεσαν το επίκεντρο της συνεισφοράς του ελεγκτικού συνεδρίου. Εμείς θέλαμε να συνεισφέρουμε για τις προτάσεις του κανονισμού και σε καμία περίπτωση δεν αναφέραμε κάτι για τις πτυχές οι οποίες αναφέρονταν διεξοδικά στο τελευταίο σχόλιο και δεν θεωρήθηκαν θετικές ενδείξεις από το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν έχουμε πείρα από ελέγχους που αναφέρονται στα νέα χρηματοδοτικά μέσα που αναφέρθηκαν. Έχουμε κάποια εμπειρία ε, όχι μέσω εκθέσεων, αλλά τυχαία εμπειρία. Ε, όταν ε, κάνουμε κάποιον έλεγχο, για παράδειγμα υπάρχει ένας συνεχιζόμενο έλεγχος ο οποίος είναι εξελίξει αυτή τη στιγμή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να περάσει από τις επιδοτήσεις τα δάνεια. Ε, μπορεί να είναι και καλή ιδέα, αλλά εμείς δεν το έχουμε ελέγξει, δεν έχουμε τέτοια εμπειρία και επομένως σε καμία περίπτωση δεν κάναμε κάποιο θετικό σχόλιο ή δεν δώσαμε μια θετική άποψη ε, επί των αλλαγών και ιδεών αυτών. Δεύτερον, αυτά τα εντελώς νέα χρηματοδοτικά μέσα εκτός ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και εκτός ευρωπαϊκής Διοίκηση. Πρόκειται για νέα ιδέα. Εμείς ως ελεγκτικό συνέδριο δεν έχουμε σχολιάσει την ιδέα αυτή, πόσο μάλλον σε λεπτομέρεια, και φυσικά δεν έχουμε και κανένα έλεγχο ο οποίος να έγινε για το θέμα αυτό. Ίσως μπορούν να προσθέσουν και κάποια πράγματα οι συνάδελφοι στα όσα είπα εγώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια. Ήθελα μόνο να πω ότι τα έγγραφα που αναφέρθηκε από τον κύριο Παρατζή έχουν ήδη αναφερθεί. Έχουν αποστελεί εκατοντάδες σελίδων με εξηγήσει. Και βέβαια ελπίζω ότι θα μπορέσουμε όλοι να συμμετάσχουμε στη συζήτηση, συνεστέφες των συναδέλφων, όλε τι πληροφορίε. Θέλω να υποβάλω όμως ε, μία ερώτηση. Αληθεύει ότι κάποιοι μισθοί δεν μπόρεσαν να καταβληθούν από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε πρόβλημα ρευστότητας. Άκουσα ότι δεν κατεβλήθησαν μισθοί. και θα ήθελα να ξέρω πόσους αφορά. Eh, Κυρία Γκρέσλε, να σα βεβαιώσω για το εξή. Εάν δεν πληρωθεί <laughs> υπάλληλο, θα το μάθετε σίγουρα και το ξέρουν όλοι. Δεν θα μπει μυστικό. μυστικό. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Κλείνουμε το σημείο 12. Στο, στο 14 έχουμε τα διάφορα. Τίποτα για τα διάφορα. Πέρα συνεδριάσεως. Και περνάμε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Χωρίς καθυστέρηση, ανακοινώνω μόνο ότι έχουμε 27 συνεδρι... Ε, Ιανουαρίου στις 9 ε, το πρωί την προσεχή συνεδρίαση. Σας ε, ενημερώνω δε ότι δυστυχώς εσάς προεδρεύω πάλι εγώ. Ο κύριος Δεμαγκίστρης είναι ασθενής. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μέχρι τις 5.30 ε, και ξαναρχίζουμε. Και κλεισμένων των θυρών έχετε υπόψη. Και κλεισμένων των θυρών οι συντονιστές. Όποιος δεν έχει θέση εδώ παρα...